Bonjour, good morning, buenos días. Καλημέρα σας σε τρεις γλώσσες. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, άρχισε η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών. Όπως είπαμε χτες, σήμερα 24 Ιουνίου, υποδεχόμαστε τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυβέρνησης της Ισπανίας, τον κύριο Φρέντο του Βαλκάβα. Τον καλωσορίζουμε. Γνωρίζετε ότι η Ισπανία αυτό τον καιρό ασκεί την ενασωμένη Προεδρία και ο κύριος Ρουμπαλκάβα προεδρεύει του Συμβουλίου Εσωτερικών και θα μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Περιλαμβάνονται θέματα όπως είναι το άσυλο, η μετανάστευση, η παράνομη, τα εξωτερικά σύνορα, η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, αστυνομική συνεργασία. Συστήμα Διαχείριση του συστήματος Schengen και ε, του σύνολο των αντιστοίχων οργανισμών για την Ευρωπόλα, ανταλλαγή πληροφοριών, ναρκωτικά, πολιτική προστασία, διευθέτηση κρίσεων και διατομιακή θεώρηση των εσωτερικών υποδέσεων. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, θα ήθελα να πω στα μέλη της Επιτροπής μας ότι εχθές στη συνεδρίαση των συντονιστών εγκρίθηκε και τυπικά η απόφαση να οριστεί ο συνάδελφός μας Αλεξάνδερ Άλβαρο της Ομάδας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών εισηγητής για το TFTP, το γνωστό SWIFT, που είναι η Διμερή Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Θα έρθει αργότερα, δυστυχώς έχει ε, ενηλυμένη υποχρέωση άλλη και δεν μπορεί να παρευρίσκεται από τις 9, θα έρθει κατά τις 10. Και θα παρακαλούσα να συζητήσουμε το θέμα αυτό από τις 10 και μετά. Να ακούσουμε πρώτα τον Υπουργό, το επόμενο τέταρτο. Θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές με τη σειρά τους για ένα πρώτο ε, γύρο ερωτήσεων. Θα απαντήσει ο υπουργό και θα ακολουθήσει γενική συζήτηση. Αλλά θα παρακαλούσα ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του SWIFT να το δούμε αργότερα. και να το συζητήσουμε από τις 10 και μετά, 10 με 11 παρουσία του εισηγητού. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός Πέρα Πέρες του Κάπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτές ε, της Επιτροπής ε, Εσωτερικών, στην οποία έρχομαι για δεύτερη φορά. Ήρθα και στην αρχή της Ισπανικής Προεδρίας, την αρχή του εξαμήνου και έρχομαι και στο τέλος. Στην αρχή ήθελα να σας παρουσιάσω τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Εσωτερικών για την Ισπανική Προεδρία και τώρα έρχομαι να σας αναφέρω τους στόχους στους οποίους φτάσαμε το εξάμεινο της Προεδρίας μας. Είχα την ευκαιρία ταυτόχρονα να έχω άτυπη συνάντηση με ορισμένα μέλη της Επιτροπής σας πριν από λίγες εβδομάδες, ακριβώς μετά τη διμερή συνάντηση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σας αναφέρω. Έρχομαι συνεπώς για τρίτη φορά ε, με ε, ορισμένους από εσά ε, συνεδρίαση και χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχω. Αν θυμάστε, στην παρουσίαση του προγράμματος εργασίας Ισπανικής Προεδρίας είχα τονίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παρούς Προεδρίας διότι ήταν η πρώτη Προεδρία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας με όλα τα σύμπαρα σε θέματα πολιτικής ασφαλείας ήταν μια προεδρία που συνέπιπτε με την έναρξη της θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Φεβρουάριο συγκεκριμένα. Είχε ήδη αρχίσει η Προεδρία. Επίσης, το Κοινοβούλιο έχει πλέον νέες αρμοδιότητες και, και νέο εκλεγέν, κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, ε, έχουμε και ε, μια νέα μορφή συνεργασίας ε, τύπου Τρόικας με τις επόμενες Προεδρίες. Αυτό συνεπαγόταν διαφορετική μέθοδο εργασίας. Η Προεδρία μας λοιπόν χρειάστηκε να εργαστεί με νέα δεδομένα, νέα ορόσημα, νέους ρόλους, ε, νέες συμπεριφορές. πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξ αυτού η δουλειά μας και πάρα πολύ ελκυστική. Όταν ξεκινάει κάτι καινούριο είναι πάρα πολύ συναρπαστικό και Είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, από τους στόχους που είχαμε θέσει και ως Προεδρία, αλλά και από τις σχέσεις που είχαμε με το Συμβούλιο, στο σύνολό του, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τις δύο χώρες ε, ε, τις οποίες συνεργαστήκαμε ε, για το τρίο. Αν θυμίστε και πάλι, όταν είχα έρθει και σας εξέθεσα τους βασικούς στόχους της Ισπανικής Προεδρίας, Θέλησα να σας πω ότι στόχος μας ήταν να αναπτυχθεί ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ακριβώς γνωρίζοντας ότι είναι πλέον κοινοτικό αυτός ο χώρος και έτσι από τη σύλληψή του έχει σχεδιαστεί και εμείς θέλαμε να ε, κατοχυρώσουμε, να εδραιώσουμε αυτό το χώρο και να αναπτύξουμε νέα στοιχεία πέρα από τα όσα είχαν αποφασιστεί πάντα υπό το φως τη Σύνθεξη Λισαβόνα. Από πολιτική απόψεω τώρα προσπαθούμε να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει υπεραξία ευρωπαϊκή και στο τομέα της ασφάλειας. Με άλλα λόγια, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί μπορούμε να προστατευόμαστε καλύτερα και στο σύνολό μας και για το καθένα ξεχωριστά. Η Προεδρία λοιπόν αυτή θέλησε κυρίως να φέρει πιο κοντά στους πολίτες τα θέματα ασφαλείας σύμφωνα με ε, το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Και από αυτό λοιπόν το γενικό πρίσμα ήταν δύο ε, διαφορετικές ε, πρωτοβουλίες, πιο στρατηγικές μεν, πιο ουσιαστικές και κάποιες άλλες πιο επιχειρησιακές, πιο λειτουργικές πιο προσανατολισμένη σε συγκεκριμένα προβλήματα στην πράξη, ιδιαίτερα αστυνομική συνεργασία. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις δύο κατηγορίες θα σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της Προεδρίας. Καταρχάς ε, να σας αναφέρω για τα πιο θεωρητικά, τα πιο στρατηγικά θέματα ε, Στη συνέχεια θα αναφερθώ στα επιχειρησιακά μέσα συνεργασίας ε, τα συγκεκριμένα για να έρθουμε και πιο κοντά στον πολίτη και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που τον απασχολούν για την ασφάλεια. Για τις στρατηγικές λοιπόν πρωτοβουλίες, η πρώτη είναι ακριβώς η έγκριση στις 25 Φεβρουαρίου μια στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας η στρατηγική αυτή είχε οριστεί από το πρόγραμμα της Στοχόλμης ήδη και προσπαθήσαμε να δώσουμε σάρκα και οστά σε ένα τμήμα του προγράμματος της Στοχόλμης. χρειαζόταν υλοποίηση και επεξήγηση το σύστημα εσωτερική ασφαλείας με τρόπο συνεκτικό, συγκεκριμένο και κατανοητό. Το σύστημα εσωτερική ασφαλείας το οποίο ε, οικοδομήσαμε τα τελευταία χρόνια. Επαναλαμβάνω, είναι απλό το έγγραφο αυτή η στρατηγική και στόχο του είναι να είναι απανάγνωστο και εύληπτο και να το χρησιμοποιούν ε, για τους πολίτες οι διάφοροι πολιτικοί θύνοντες. Η στρατηγική μας λοιπόν ε, περιέχει τέσσερα βασικά στοιχεία. Πρώτον, περιέγραψε τους στόχους και τις κοινέ απειλές. Απειλές που γνωρίζουν όλες οι χώρες και είναι κοινέ και πάρα πολύ γνωστές. Το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, το έγκλημα στο κυβερνό χώρο, ε, διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Είναι κοινέ λοιπόν αυτές οι απειλές, τις οποίες περιγράφουμε. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα της στρατηγικής ασφαλείας. Ακολουθεί η περιγραφή του μοντέλου εσωτερικής ασφάλειας που οικοδομούμε σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια με διάφορα ε, όργανα, ε, οργανισμούς, Europol, Eurojust κτλ. Τρίτον, στρατηγική πάντα για τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάντα διέπουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέναντι σε αυτούς τους κοινούς κινδύνους και απειλές είναι αδιαπραγμάτευτα τα στοιχεία, αναπαλωτρίωτα και ίδια η βάση και η ουσία της Ένωσης. Κράτος δικαίου, δηλαδή προστασία των δημοσίων ευθυριών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διαφάνεια, ευθύνη ε, στη δημόσια δράση, συμπερίληψη, ε, ανεκτικότητα, βεβαίως σεβασμός της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών. Όλα αυτά είναι αρχές και αξίες που αποτελούν θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να είναι και τμήματα της στρατηγικής ιστορικής ασφάλειας. Και τέταρτον, χαράζουμε δέκα ε, γραμμές ε, κοινή συνεργασίας αστυνομικής και δικαστικής ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που στην αρχή περιγράφουμε. Οι γραμμές αυτές λαμβάνουν κυρίως υπόψη την ανάγκη αναθεώρησης, ε, ενημέρωσης Γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει σήμερα το οργανωμένο Διεθνέ έγκλημα είναι η δυνατότητα που έχει να μεταλλάσσεται, να εξελίσσεται, να αλλάζει. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να προσαρμόζουμε τη δράση μας με ε, κοινά ε, μέσα και εργαλεία εργασία. Βεβαίως χρησιμοποιούμε και νέες τεχνολογίες και ε, τις υπηρεσίες πληροφοριών. Η πληροφορία είναι βασικότατο στοιχείο ε, των εργασιών μας για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους ακριβώς που έχουμε ενώπιόν μας. Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα. Σήμερα έχουμε στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας, επαναλαμβάνω, η οποία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και ε, ενέκρινε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνέχεια. Εκτός λοιπόν από αυτές τις πιο ουσιαστικές αποφάσεις ε, θέσαμε σε λειτουργία και την Επιτροπή Κώση εσωτερική ασφάλεια δηλαδή. Είναι μια νέα επιτροπή η οποία ιδρύεται από τη Συνδίκη τη Λισαβόνα. Και όπω είχα την ευκαιρία να σα εξηγήσω την προηγούμενη φορά που ήρθα, την πρώτη φορά, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε άλλον έναν οργανισμό, όχι. Αλλά έναν οργανισμό χρήσιμο που να αντικαταστήσει ορισμένου που σήμερα υπάρχουν αλλά έχουν αποδείξει στην πράξη ότι δεν λειτουργούν σωστά. Για παράδειγμα, η Task Force, η ομάδα εργασίας των επικεφαλής ε, των αστυνομιών που δεν λειτουργήσε καλά όπως είχαμε φανταστεί. η Επιτροπή λοιπόν αυτή της εσωτερικής ασφαλείας αντικαθιστά ορισμένα όργανα που σήμερα υπάρχουν ε, και είναι ένα όργανο αστυνομικής συνεργασίας πάρα πολύ σημαντικό. Συστήθηκε λοιπόν η Επιτροπή αυτή, συνήλθε και ε, έχει ήδη ε, προχωρήσει σε κάποιες αποφάσεις σημαντικές. Για παράδειγμα, μέσω ενός εγγράφου το οποίο εκπώνησε στο εσωτερικό της η Επίτροπη αυτή με ε, τους οργανισμούς Europol, Eurojust, Frontex κυρίως. Ένα έγγραφο λοιπόν το οποίο επέτρεψε στο Συμβούλιο να κάνει μια συζήτηση για την εσωτερική ασφάλεια και το Πού βρίσκεται, ποια κατάσταση επικρατεί σήμερα τον Ιούνιο βάσει ακριβώ αυτού του εγγράφου που ε, προετοίμασε η Επιτροπή Εσωτερική Ασφάλειας. Πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη αυτή η ε, συνεδρίαση. Αποφάσισε το ε, Συμβούλιο αυτό να γίνεται κάθε χρόνο πάντα βάσει εγγράφου που θα εκπονεί η Επιτροπή εσωτερική ασφάλεια. σε συνεργασία με τους διαφόρους οργανισμούς. Η Επιτροπή εσωτερική Ασφάλειας είναι το σημείο αναφορά και συγκεντρώνει ε, αυτούς τους οργανισμούς Europol, Eurojust, Frontex κλπ. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα όργανο κάπου να συνέρχονται, να συνεδριάζουν μαζί, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να βελτιώνουν τους μηχανισμούς συντονισμού. Αυτό γίνεται λοιπόν ήδη σε επιχειρησιακό επίπεδο και έχουν γίνει κοινέ αστυνομικέ επιχειρήσεις πολύ σημαντικές και σιγά σιγά θα ε, ενισχύσουν την κοινή μας προσπάθεια στην ασφάλεια και στην άμεση ασφαλείας. Έχουμε λοιπόν αυτή την επιτροπή με συγκεκριμένους στόχους που καλείται να αντικαταστήσει ορισμένες επιτροπές που δεν λειτουργήσαν σωστά και χρειάζονται αντικατάσταση. Στη συνέχεια, Όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εγκρίναμε στο τελευταίο Συμβούλιο Ιστορικών και Δικαιοσύνης τη θέση σε ισχύ του προγράμματος δράσης ε, της Στοκχόλμης. Σε χρόνο ρικόρ έγινε αυτό και θα πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια. Θα έχω την ευκαιρία να το κάνω επανειλημμένα σήμερα το πρωί. Ε, την εξαιρετική ε, δουλειά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, αρχίσουν να λειτουργούν αυτές ε, οι δράσεις. Και στο πρόγραμμα της Σοχόλμης λοιπόν έχουμε δράσεις με προτεραιότητες, με ε, κατανομή ευθυνών, ανάθεση ευθυνών και χρονοδιαγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να αναπτυχθεί η συνεργασία μας που είναι ακριβώς αυτό το πρόγραμμα της ΟΧΟΛΜΗΣ... το οποίο αποτελεί τον κύριο άξονα ε, ασφαλείας στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, σύμφωνο ε, μετανάστευση και άσυλο. Ε, νομίζω ότι η αρμόδια υφυπουργό ήρθε χθε στην Επιτροπή σας και είχατε την ευκαιρία να το συζητήσετε. Δεν θα επεκταθώ εγώ σε αυτό. Απλώς να θυμίσουμε ότι το σύμφωνο αυτό είναι το έμβριο μια πρώτη προσπάθεια κοινή ε, πολιτικής στο άσυλο και τη μετανάστευση και χαράξαμε τις ε, κατευθύνες γραμμές για την εργασία των επόμενων ετών για να εντρεωθεί μια κοινή πολιτική μετανάστευση και ασύλου όπως ορίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και το πρόγραμμα της Στοχόλμη. για την νόμιμη μετανάστευση, η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, Τη διακίνηση ανθρώπων, προστασία των συνόρων, συνεργασία με τρίτε χώρες και όλες τις διαδικασίες συνολικής αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ρευμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Στη συνέχεια επεξεργαστήκαμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Την πρώτη φορά που ήρθα εδώ σας είπα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το θέμα. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης καθυστέρησε ε, τη θέση ισχύ αυτού του συστήματος, στην παρέτηνε μέχρι το 2013 την προπαρασκευαστική περίοδο. Δηλαδή είναι περίπλοκο το θέμα με διαφορετικές ευαισθησίες στα κράτη-μέλη που δυστυχώς ε, οι θέσεις τους απέχουν πολύ. Υπάρχει Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξη στο Άσυλο. Είχα την ευκαιρία να υπογράψω τον αντίστοιχο κανονισμό μαζί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου πριν από λίγε εβδομάδε. Το γραφείο αυτό θα συγκεντρώσει την εμπειρία μας για το άσυλο και θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα λόγω πληθώρας ε, αιτήσεων ασύλου δεν μπορούν να ανταποκριθούν ε, σε όλο αυτό τον όγκο. Και επίσης έχουμε εργαστεί σε διάφορα θέματα, οδηγίες και κανονισμούς που μας κληροδότησε η Σουηδική ε, Προεδρία Δουβλίνο, Eurodac και οδηγίες για υποδοχή και επανεγκατάσταση που φαντάζομαι ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υλοποιηθεί όταν τα τρία θεσμικά όργανα θα έχουν συμφωνήσει. Για να βρούμε τα καλύτερα δυνατά νομικά μέσα για να τα θέσουμε όλα αυτά σε ίσχυ. Επίσης προχωρήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Σύλλου αν και θα πρέπει κανείς να αναγνωρίσει ότι είναι πιο αργά τα βήματα πρόοδου από εκείνα που περιμέναμε, γιατί είναι τεράστιες οι δυσκολίες και πάρα πολύ δύσκολο επίσης να ξεπεραστούν θέσαμε σε ισχύ τον κανονισμό του Frontex και πάλι θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσει το Συμβούλιο να ασχοληθεί με αυτό το αρχικό κείμενο και να το διεκπαιρεώσει. Στις 24 Φεβρουαρίου ήδη κατέθεσε πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε ο κανονισμός αυτός ασχολείται με την ενίσχυση του ρόλου του Frontex βάσει της εμπειρίας που έχουμε και μεταξύ άλλων να έχει ε, εκείνα τα στοιχεία ε, και τα μέσα που χρειάζεται το Frontex για να λειτουργήσει σωστά. Και για τους ετούντες άσυλο επίσης θέλουμε ε, ένα τέτοιο οργανισμό να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των ετούντων κτλ. Λοιπόν, ο κανονισμός εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση έχει λίγα χρόνια ζωής και λειτουργίας ο Frontex, αλλά έχει τεράστια αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του. Τώρα βρισκόμαστε σε δεύτερη ανάγνωση και ελπίζω να δώσει το οριστικό και η Βελγική Προεδρία. Επίσης, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κάναμε βήματα προόδου στα συστήματα SIS-2 και VIS, ειδικά το SIS-2, το σύστημα ε, ε πληροφόρηση στο Σέγγεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν και περίπλοκο, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρώπη. Πάντα θα πρέπει να συνοδεύεται ε, αυτό από τις απαραίτητες εγγύσεις για την ασφάλεια. Ξέρω ότι είναι το θέμα δύσκολο. Από πλευράς τεχνολογικής υπήρχαν διάφορες εξελίξεις. Το 2009 το Συμβούλιο, τον Ιούνιο αν δεν απατώμε, είχε πάρει κάποιες αποφάσεις. Ε, εκεί εργαστήκαμε και συντονίσαμε ε, τη θέση σε ισχύ των αποφάσεων βάσει ε, προηγουμένων εμπειριών για το ΣΥΣ2. Δώσαμε ε, την έγκρισή μας για το πρώτο ορόσημο που είχαμε θέσει ε, το 2009. Νομίζω ότι προχωρούμε έτσι με λογικούς ρυθμούς και το δεύτερο ορόσημο ελπίζω σύντομα να επιτευχθεί και να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες το ΣΥΣ 2 σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν προβλεφθεί και το χρονοδιάγραμμα. Και το ΒΙΣ επίσης. Για το SWIFT, το TFTP, πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδότησης τρομοκρατίας, είπε ο πρόεδρος... Α, έχει φτάσει ο εισηγητής. Ωραία. Μπορούμε να το συζητήσουμε επί της ουσίας. Πρέπει να σας πω μόνο ότι η Ισπανική Προεδρία το κληρονόμησε αυτό το θέμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς ε, άλλωστε την όλη εξέλιξη και προϊστορία και πώς το Κοινοβούλιο απέριψε την ε, ενδιάμεση συμφωνία και επειδή ήταν κατεπήγον το θέμα και έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρξει νέα συμφωνία γιατί και η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κομισιόν και το Συμβούλιο ήμασταν πεπισμένοι ότι είναι καλό εργαλείο ενίσχυση της συνεργασίας μας. Ε, επιταχύναμε λοιπόν για να εργαστούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Λάβαμε υπόψη τις ε, προτάσεις του Κοινοβουλίου, τις επικρίσεις επίση του Κοινοβουλίου ε, στην προηγούμενη προσωρινή συμφωνία. Και επίση πρέπει να, να, να σημειωθεί και η αντίσταση, η διαφωνία των ΗΠΑ. Ε, νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, υπήρξε και ψήφισμα του Κοινοβουλίου, εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο πριν εγκριθεί η εντολή και με αυτά τα δύο στοιχεία αναφοράς το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην εκπόνηση μια νέα εντολή και είμαστε στα τελευταία στάδια. Χωρίς να προεξοφλήσω τη συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι η νέα συμφωνία αυτή που έχουμε ενώπιόν μας λαμβάνει υπόψη σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, λαμβάνει υπόψη επίσης και τις προβλέψεις της εντολής και μάλιστα με μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ πιστά για να μεταφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα τις θέσεις και των κρατών μελών και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί ξέρετε και τα κράτη-μέλη δεν ταυτίζονται πάντα στις απόψεις τους. Γενικά νομίζω ότι η συμφωνία είναι πάρα πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Συμπεριλαμβάνει τις βασικές προτάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την εντολή και έτσι κι θα συζητηθεί Μέχρι χτες το Συμβούλιο αναθεωρούσε μερικά στοιχεία ε, για να ε, υλοποιήσει τα όσα ζητάει το Κοινοβούλιο και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί ε, ξεκίνησε η γραπτή διαδικασία για να μπορέσει να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες η συμφωνία και να ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι πίεζε ο χρόνο, γι' αυτό και δράσαμε πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω θα πρέπει να, να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα που υπάρχει αυτόν τον καιρό γιατί δημιουργεί και ανασφάλεια. Να ξεφύγουμε από αυτή την αβεβαιότητα και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν άψογη στις διαπραγματεύσεις. Τελειώνω με αυτέ τι πιο στρατηγικέ ε, πρωτοβουλίε ε, Αναφέρω με ε, στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις διατλαντικές σχέσεις, γνωρίζετε ότι σήμερα τα θέματα ασφαλείας είναι κυρίως θέματα εσωτερικής πολιτικής, αλλά και εξωτερικής ταυτόχρονα. Και είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο να έχουμε συμφωνίες με χώρες που αντιμετωπίζουν απειλές και κάποιες άλλες που μπορεί να μην αντιμετωπίζουν ακριβώς σήμερα απειλές, αλλά μπορεί να χρειάζεται διάλογος και διαπραγμάτευση μαζί του. Γιατί είτε από εκεί προέρχονται οι ε, απειλές είτε είναι χώρες διέλευσης. σε αυτές τις εξωτερικές σχέσεις είναι σημαντικές ε, σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, θελήσαμε να τις ε, βελτιώσουμε. Σας μίλησα για το SWIFT που είναι μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ανταλλάξαμε απόψη για τη διεθνή τρομοκρατία στο Τολέδο σε ένα άτυπο συμβούλιο. Πάρα πολύ σημαντική ήταν η ανταλλαγή απόψεων και προέκυψε μια κοινή δήλωση που μας υποχρεώνει να εργαστούμε στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας γιατί είναι βασικός στόχος της διεθνούς τρομοκρατίας ακόμα αυτό, έγινε μια σύνοδος κορυφής πάρα πολύ σημαντική και είχα την ευκαιρία να σας αναφέρω εδώ και ε, υπογράψαμε και κοινή δήλωση για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας που είναι πάρα πολύ σημαντική και δείχνει ποιες είναι οι διάφορες σχέσεις που έχει η Ευρώπη με τις Ηνωμένε Πολιτείες και πώς αντιμετωπίζει αυτό το νέο είδος τρομοκρατίας. Η νέα κυβέρνηση στις Ηνωμένε Πολιτείες βοήθησε να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες που είχαμε για την αντιτρομοκρατική μας δράση. Σήμερα ταυτιζόμαστε πλήρως με τις Ηνωμένε Πολιτείες, τις αρχές, τους στόχους και τις αξίες μας και αυτό μας επέτρεψε να υπογράψουμε μια συμφωνία πάρα πολύ ουσιαστική. που διατρανώνει και την αποφασιστικότητα και της Ένωσης και τον ΗΠΑ απέναντι σε μια τρομοκρατία που αφισβητεί τη δημοκρατία μας, τον τρόπο ζωή μας και γνωρίζει όμως και ε, η ε, συμφωνία εκτός από την αποφασιστικότητα ότι είμαστε δημοκράτες, ότι είμαστε ανεκτικοί και υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι και μορφές ε, ζωής και κοινωνικής. Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν από πολιτική πλευρά, γιατί όπω γνωρίζετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Δικαστήρια, αστυνομία, ε, μυστικέ υπηρεσίε, αλλά και πολιτικέ δηλώσει. Να λέμε ποια είναι η θέση μα στον κόσμο. Είμαστε και αποφασιστικοί και ανεκτικοί. Έχουμε και πυγμή και ανοχή. Τώρα έχουμε τις ε, πρωτοβουλία στη δεύτερη δέσμη αυτών, γιατί έτσι έγινε η διαίρεση των ενεργειών μας. Έχουμε αυτή την συνεργασία όπου δουλέψαμε μέσα από συγκεκριμένες συζητήσεις αλλά και συμπεράσματα προέβημενη στην έγκριση κάποιων εγγράφων και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη προς τις διοκτικές ε, αρχές ε, ε, γιατί ακριβώς είπαμε ότι η συνεργασία είναι καλύτερη όταν υπάρχει ε, εμπιστοσύνη, αμοιβαία. Ε, και από την άλλη μεριά, όσο πιο καλά συνεργάζεται κανείς, χτίζεται η εμπιστοσύνη και ε, μετά στη συνέχεια γίνεται κανείς πιο αποτελεσματικός. Πάνω σε αυτό τον άξονα επομένως προχωρήσαμε στην αστυνομική συνεργασία ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποιες κοινέ ομάδες συνεργασίας με διμερείς μηχανισμούς, με κάποια συμφωνία τύπου ε, που ενεκρίθηκε, χρησιμοποίησε η Προεδρία με όλες τις χώρες και έτσι θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ανταλλαγής για την κατάρτιση των αστυνομικών, κάτι σαν το έρασμος αλλά για τους ε, αστυνομικούς. Και έτσι να βελτιώσουμε την μετώπιση της εγκληματικότητας και το σχετικό δίκτυο. Είπαμε έτσι να αξιοποιήσουμε κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου για κάποιες πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις αθλητικές και πολιτιστικές. Ό,τι τέλος πάντων καλύπτει η αστυνομική συνεργασία. Επίση ασχοληθήκαμε με την πρόληψη αλλά και καταστολή της τρομοκρατίας. Διευκολύναμε τις ε, ανταλλαγέ μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Έτσι είχαμε καλύτερη συνεργασία. Ασφάλεια σε σχέση με τις εκρηκτικές ύλες ομάδες συνεργασίας με τρίτες χώρες για καταπολέμηση τέτοιου είδους τρομοκρατίας. Επίσης επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας όσον αφορά το να αναζητηθούν πόροι, οι πόροι αυτοί που ξεπλένουν οι εγκληματικέ οργανώσεις μέσα από παράνομες ενέργειες. Οπότε βοηθήσαμε στο να έχουμε κάποιες υπηρεσίες για να παρακολουθούν αυτές τις ε, ενέργειες για το ξέπλυμα του χρήματος του οργανωμένου εγκλήματος επίσης. Χαράξαμε μια στρατηγική για να καταπολεμήσουμε στην Δυτική Αφρική το οργανωμένο έγκλημα, καταπολέμηση των ναρκωτικών, γιατί ξεκινήσαμε από το ότι η κοκαίνη μπαίνει στην Ευρώπη από τη Δυτική Ευρώπη και η ηρωίνη από την Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε επομένω αυτές τις ε, δύο διαδρομές, προσπαθήσαμε να τις μπλοκάρουμε. Και έτσι ο καθένας έκανε ό,τι θεωρήθηκε εξειδικεύσή του. Επίσης καταπολεμήσαμε το δουλεμπόριο ανθρωπίνων ζώων και ε, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιους ε, συνδέσμους για συνεργασία το έγκλημα κατά του περιβάλλοντος καθώς και τα τοξικά απόβλητα. Λαθρομετανάστευση, έλεγχος των συνόρων. Και ακριβώς γι' αυτό θεσπίστηκαν 29 μέτρα, μια ολόκληρη δέσμη, ούτως ώστε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ε, αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία που σας προανέφερα. Προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται με τις ε, νέες τεχνολογίες όσον αφορά την είσοδο στην Ευρώπη για να μπορούμε να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των Ευρωπαίων μέσα στην Ένωση και έτσι με την πρόοδο της τεχνολογίας να γίνει η ζωή πιο εύκολη. Επίσης ε, διάφορους, ε, διάφορες υπηρεσίες για την φύλαξη των συνόρων. Πλαισίωση των θυμάτων του εγκλήματος και συγκεκριμένα της ε, τρομοκρατίας, οδική ασφάλεια, ανταλλαγή πληροφοριών, ε, ανταλλαγή επίσης ε, πληροφοριών για το σοφρονιστικό σύστημα, και προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τι ε, απειλέ που από κοινό αντιμετωπίζουμε. Επίση, ε, χαράξαμε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα σαν ε, Ευρωπαϊκή Προεδρία που θεωρήσαμε ότι καταρχήν ο απολογισμό είναι ικανοποιητικό σε σχέση με όσου έχουμε πετύχει και επίση μια που έχω το βήμα θα πρέπει για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Ε, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Μα βοήθησαν πάρα πολύ να υλοποιήσουν το πρόγραμμά μα σε όλα τα κρατημέλη Επίσης βοήθησαν και οι υπηρεσίες του Συμβουλίου, αλλά και οι ευρωβουλευτές οι οποίοι βοήθησαν, συζήτησαν ε, και συνέβαλαν στο να χαράξουν αυτούς τους άξονες ε, πάνω στις οποίες κινήθηκε το ρόλο της Προεδρίας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτόν τον ε, απολογισμό του εξάμεινου της Προεδρίας όσον αφορά δικαιοσύνη και εσωτερικά. Τώρα θα προχωρήσουμε σε έναν πρώτο γύρο τραπέζης, ούτως ώστε να ακούσουμε ερωτήσει απαντήσει από όλε τι πολιτικέ πτέρυγε του Κοινοβουλίου. Πρώτα-πρώτα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει το λόγο ο κ. Δία Δεμέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Υπουργό που ήρθε για να μας κάνει αυτή την τόσο πλήρη σύνοψη των όσων επιτέλεσε η Γερμανική Προεδρία στα θέματα δικαιοσύνης εσωτερικών. Τζάι. Έχω κάποιες ε, επικρίσεις, όχι πάρα πολλέ όμως κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το έργο σας. Πρώτα-πρώτα κάποιες ερωτήσεις, διότι παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας ε, αναφέρατε όσον αφορά ε, το επιχειρησιακό, το στατηγικό περιεχόμενο της διαδρομής της Προεδρίας. Συμφωνώ στα όσα μας αναφέρατε γιατί ήταν πάρα πολύ πλήρη αυτό που μας είπατε. Τώρα, πιο συγκεκριμένα κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το άσυλο. Σημειώθηκε πρόοδο σε συγκεκριμένα θέματα όπως η δημιουργία της σχετικής υπηρεσίας αλλά και αυτό το νέο ταμείο για τους πρόσφυγες. Από την άλλη μεριά όμως ακούσαμε τι είπατε όσον αφορά τις δυσκολίες του κοινού συστήματος χορήγησης άσυλου και έχουμε την τροποποίηση των σχετικών ομοθετημάτων κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αντίθετα έχει εμπλακεί. Τι έγινε με την ολοκλήρωση τη δέσμη μέτρων για το άσυλο. Τώρα τι γίνεται με τα εξωτερικά σύνορα. Η έγκριση αυτού του προγράμματος και των σχετικών μέτρων όσον αφορά τους ανήλικους τους ασυνόδευτους είναι κάτι που δεν μας αναφέρατε. Όπως και το προηγούμενο θέμα, δεν μας είπατε τίποτα. Τι γίνεται, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, όσον αφορά την καταπολέμηση της λάθρομετανάστευσης, θα πρέπει να προχωρήσουμε συνάπτοντας συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως το Μαρόκο. Ή θα πρέπει να πλησιαστούμε περαιτέρω τις υπάρχουσες συμφωνίες. Επίσης και όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα, όπως συζητήσαμε και χθε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει το 2013, τι θα γίνει με τον νέο κανονισμό της Frontex. Μας τα είπατε, αλλά σε πολύ γενικές γραμμές. Θέλουμε πιο συγκεκριμένα να μάθουμε ακριβώς τι θα γίνει με την ΚΝΟΥΡ του Διεθνούς Φορέα για τους πρόσφυγες. Τώρα, όσον αφορά το SWIFT, ήρθατε και μας είπατε στην Ολομέλεια ε, τα του απολογισμού της Προεδρίας. Και ξέρετε ότι έρθει η ώρα να ψηφίσουν οι Ισπανοί, συνάδελφοι της Ισπανικής συνιστώσεις, κάποιοι απέσχον και άλλοι ψήφισαν υπέρ. Τι γίνεται όμως, αυτό θα πρέπει να το ρυθμίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε γιατί θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να κληθεί ο καθένα να πάρει τη θέση του, γιατί μέσα στη δημοκρατία θα πρέπει να, να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι καθαροί και ποιοι όχι. Και αυτό ακριβώς αφορά και το, όσα γίνονται και στις ΗΠΑ. Έχουμε επίση το κείμενο για το οποίο είναι υπεύθυνο ο κύριο Άλβαρο και τώρα όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία Έχουμε συνεργασία, αλλά δεν την έχουμε στα θέματα της αστυνομικής έρευνας. Ε, για το οργανωμένο έγκλημα σημειώθηκε πρόοδος, είχαμε το συμβόλαιο της 4ης Ιουνίου και έγινε μια πρώτη παρουσίαση για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για καταπολέμηση των ναρκωτικών και καταπολέμηση συγκεκριμένα ηρωίνης και κοκαίνης. Τώρα όσον αφορά το έγκλημα ε, στον κυβερνοχώρο. Συγγνώμη να με συμπαθούν οι διερμηνεί γιατί τα λέω πάρα πολύ γρήγορα. Επομένω, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά την ε, παιδεραστία και όσον αφορά αυτό το κυβέρνο έγκλημα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Επίση, θα πρέπει να δούμε πώ θα καταπολεμήσουμε την ε, πλαστογράφηση του ευρώ και εν κατακλείδη κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Για πετε μας για την Europol. Στη Στοκχόλμη είχε προβλεφθεί να κατέβει σχέδιο κανονισμού για την Europol μέχρι το 2013. Σύμφωνα με τόσο ορίζει η συνδικητή της Μήπω Μήπως κύριε Πρόεδρε θα μπορούσατε να μας πείτε εάν αυτός ο κανονισμός θα προβλέπει νέες αρμοδιότητες για την Europol ή απλώς θα αφορά ε, την, τα όσα προβλέπει το άρθρο 88 της συνθήκης. και επαναλαμβάνω ότι στα περισσότερα συμφωνήσαμε, σε κάποια διαφωνήσαμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα δικαιοσύνη. Τώρα ε, πρέπει να δώσουμε σε όλου ε, το λόγο. Ε, φυσικά και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, όμω λάβετε υπόψη το χρονικό περιορισμό. Γιατί θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο συνοπτικοί. Γιατί θα πρέπει να προλάβουν να μιλήσουν και οι συντονιστέ. Και τώρα, ε, κύριος Μωράης για το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ευχαριστώ. Θα είναι δύσκολο να είμαι σύντομος ε, γιατί έχουμε και τα θέματα TFTP. Θα αρχίσω με το βασικό θέμα. Θέλω να πω στον Υπουργό ότι οι σοσιαλιστές πιστε... αναγνωρίζουν Συγγνώμη, Κλοντ, υπάρχει ένα θέμα με τη μετάφραση, ένα λεπτάκι. Uh, Μπορείτε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Α, να, αντλήσω και το δίδαγμα ότι πρέπει να συνεχίσω τα μαθήματα Ισπανικών. Uh, ε, Υπουργέ, πρώτα απ' όλα, η πολιτική μας ομάδα δεν θεωρεί ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα, ε, δηλαδή ότι έκανε ιδιαίτερε προσπάθειες στον τομέα Τζάι η Ισπανική Προεδρία. Πριν περάσω το TFTP ήθελα να πω Βέβαια ότι ε, υπήρξαν σημαντικές νίκες γιατί δεν ήταν και εύκολη η Προεδρία. Παραδείγματος χάρη για τους υπόπτους, διαδικαστικά έγκαια. Ήταν ένα θέμα που είχε θαυτεί ε, πριν από την Προεδρία ε, της Ισπανίας. Ε, τώρα έχουμε τις μεταφράσεις, είναι προτεραιότητα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Υπήρξαν διάφορα μηνύματα που κατέδειξαν ότι είναι αποφασισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προοδεύσει σε ζητήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το αναγνωρίζουμε αυτό. Δεύτερον, ε, μέσα στο πρόγραμμα της Στοχόλμης υπάρχει πλέον ένα σχέδιο δράσης, ένας οδικός χάρτης. Ε, όταν ε, συστάθηκε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ουσιαστικά είχε τα πάντα μέσα. Όλοι κάτι μπορούσαν να βρουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και χρειαζόμασταν τον οδικό χάρτη. Τώρα έχουμε σχέδιο δράση, έχουμε και χρονοδιάγραμμα. Στην Ολομέλεια βέβαια είχαμε θέματα εμείς για την παράνομη μετανάστευση και άλλα ζητήματα που θέλαμε ε, να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Τέλος πάντων, καλό είναι που έχουμε πλέον ε, το νοδικό χάρτη. Αναγνωρίζουμε ε, κάποιες επιτυχίες, αλλά υπολείπονται ζητήματα που μας ανησυχούν. Κάποια οριζόντια ζητήματα πρώτα απ' όλα. Τα προβλήματα στον τομέα J με τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Πώς θα λύσετε αυτό το θεσμικό ζήτημα τηρώντα το πνεύμα της συνθήκης. Ε, είμαστε συνομοθέτες εδώ στο Κοινοβούλιο και είναι θέμα ύψης της προτεραιότητας για την ομάδα μου. Δεύτερον, η, αυτή η διχοτόμηση στι γενικές διευθύνσει είναι γενικό πρόβλημα. Ε, Πώ τι θα γίνει στον τομέα Τζάι με αυτή τη διχοτόμηση. Έχουμε δύο διαφορετικού, δύο συναρμόδιου επιτρόπου Μπορεί να μην θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, αλλά τουλάχιστον εγώ το θέτω, εφόσον πλησιάζεται και στο τέλος της Προεδρίας, για το πακέτο ασύλου, ε, να καταγράψετε μια ανησυχία που έχουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Δεν θέλαμε να χωριστεί στα δύο αυτό το πακέτο του ασύλου. Υπάρχει το Γραφείο Υποστήριξη Ασύλου για την επανεγκατάσταση, ε, της άλλα ζητήματα, τώρα έχουμε τα διαδικαστικά, θα, τα, θα τα αναφέρουν και άλλοι συνάδελφοι. Το πρόβλημα είναι ότι άμα ε, χωρίσουμε το πακέτο θα δημιουργήσουμε αντιδικίες. Ε, το συστήσαμε και με την Επίτροπο Μάλμστρομ, αλλά ξέρουμε το περιεχόμενο είναι αυτό που έχει σημαντικό και το, στο Συμβούλιο προκύπτουν τα προβλήματα θα θέλαμε να μας πείτε κατά τη γνώμη σας πώς θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες ε, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και πώς θα ε, διατηρήσουμε τη συνοχή του πακέτου. Θα σταματήσω τώρα γιατί μου ζήτησε ο Πρόεδρος να είμαι σύντομος. Για το TFTP, Πρόεδρε, ε, πώς ακριβώς θέλετε να γίνει συζήτηση, να σχολιάσω τώρα το TFTP ή θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή. Νομίζω ήρθε η ώρα, περιμέναμε τον κύριο Άλβαρο όλοι. Ήρθε. Οπότε, ναι, σχολιάστε και τα ζητήματα του FTP. Μάλιστα και υπόσχομαι θα είμαι σύντομο. Ε, η πολιτική μας ομάδα έχει σαφή άποψη. Μετά την αρνητική ψήφο το Φεβρουάριο, σημειώθηκαν διάφορες θετικές εξελίξεις Συμφωνία Πρόσβαση στα δεδομένα επικύρωση, διαγραφή, ε, ε, με επανόρθωση, με μη διακριτική μεταχείριση. Βελτιώθηκε πολύ η συμφωνία. Ε, σαφώς όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θέλουν να συμπεριληφθούν συμφωνία. Εν συντομία, όλοι τα γνωρίζουν, έτσι. Εμείς τουλάχιστον ζητήσαμε παρακολούθηση και διαφύλαξη των δεδομένων άρθρο 12. Θέλουμε να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Έκανε κάποια βήματα η Ισπανική Προεδρία γι' αυτό. Επίσης, τι άλλο ζητήσαμε. Ε, για να εμφανιστούν στις δηλώσεις της συμφωνίας τη FTP. Δεν θα σας τα απαριθμίσω, δηλαδή αναφορά στη Γενική Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων, οι ομάδες δεδομένων, ε, η χρήση από τη Europol. Δεν έχουν ρυθμιστεί όλα αυτά τα ζητήματα και πιστεύουμε πως ε, η Προεδρία έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες, αλλά σαφώς ε, υπάρχουν ακόμη ανησυχίες ε, για την ε, συλλογή δεδομένων στην επικράτεια της Ένωσης, το θέμα του χρονισμού. Συμφωνούμε με τον εισηγητή που επιμένει για τα τρία χρόνια. Αλλά περιμένουμε τώρα, θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθεί ε, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες των διαπραγματεύσεων. Να γνωρίζουμε λοιπόν ε, τη σημειωθήσα πρόοδο, να γνωρίζουμε τι προσπάθειε τη Προεδρία για να ανοίξει ε, τη συμφωνία και να συμπεριληφθούν και άλλα σημεία. Τώρα είμαστε στι τελευταίε ημέρε, πλησιάζουν στο τέλο οι διαπραγματεύσει, θα δούμε. Ευχαριστώ για του φιλελευθέρου, του κύριο Άλβαρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich das Δεν νομίζω για βάλτε τίποτα ακουστικά, συνάδελφοι, περιμένω. Καλώς. Ε, ε, νομίζω δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπε ο Κλοντ Μωράες. Ε, τόνισε ποιες είναι οι πρόοδοι για μας. Ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το πώς έχει σήμερα η κατάσταση των πραγμάτων. Όταν μιλήσατε για τα προγράμματα, αναφέρατε τις δύο λέξεις. Εμπιστοσύνη και κάτι άλλο που ακούω πολύ συχνά από τον Επίτροπο και το Συμβούλιο αδύνατο. Ε, πώς γίνεται αυτό τώρα. Ε, ανοιχτές πολλές ερμηνείες, να δούμε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Εχθές, συνεδρίαση Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Θα μπει ένα άρθρο που ζητάει το Κοινοβούλιο στην απόφαση του Συμβουλίου για να είναι δεσμευτικά αυτά δηλαδή τα ευρωπαϊκά στοιχεία να αξιολογούνται ε, στην επικράτεια της Ένωσης, όχι να πηγαίνουν χίδι στις Ηνωμένε Πολιτείε, το περίφημο bulk transfer. Και μέσω πρόθεσμα οι συντονιστές θεωρούν το, ε, ε, ότι πρέπει ε, να ε, είναι τριετία το μεσοπρόθεσμο και ζητήσαμε και από τον πρόεδρό μας εχθές να κάνει επιστολή. Εχθές το βράδυ, 11.30 ώρα παρακαλώ, με πήρε η Ισπανική Προεδρία τηλέφωνο από τη Μαδρίτη. Ε, αργά δεν είναι. Γιατί εγώ είχα ραντεβού στις 7 το απόγευμα ε, με τον πρέσβη σας, ο οποίος με αγνόησε. Και κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση του Κορεπέρ ήμουν στη διάθεσή του όλη την ημέρα αν υπήρχαν προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκανε. Α πούμε, θέλανε να με πάρουν τηλέφωνο να το συζητήσουμε γιατί στι 11.30. Αυτή η τριετία, από ό,τι φαίνεται τώρα, έχει γίνει το ζήτημα κλειδί και γόρδιος δεσμός και λέει, θεωρούν ότι εμείς βάλαμε νέα εμπόδια και νέα θέματα. Μα από τη Δευτέρα τουλάχιστον το γνωρίζει η Προεδρία ότι μιλάμε εμείς για τριετία. Την Τρίτη Επίσης το κοινοποίησα στην ερχόμενη Προεδρία ε, στο Βέλγιο ε, γραπτός και με διαβεβαίωσαν ότι θα το διαβιβάσουν στο Κορεπέρ, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το μπλόκαρε η Ισπανική Προεδρία. Εχθές μάθαμε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ότι καμία χώρα εκτός από τη δική μου δεν είναι πρόθυμη να υποστηρίξει την τριετή αυτή και πρέπει να σας πω ότι η δική μας πρόταση έχει ε, μετριαστεί, γιατί εμείς ζητούσαν με βάση του άρθρου 1 εδάφιο 2 αυτόματη καταγγελία αναστολή της συμφωνίας, αν δεν γινόταν αυτό. Ε, εμείς βάλαμε νερό στο κρασί μας και με πολύ βαριά καρδιά δεχτήκαμε τελικά το σάλκο Σίντερ του review και όχι αυτόματα, που είναι απλώς δήλωση προθέσεων θα δείξει ενδεχομένω και να το επανεξετάσουμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πιο ε, απαλή διατύπωση. Κάτι που με εξέπληξε ήταν ότι πολλοί μας λέγανε ότι είναι αδύνατη αυτή η τριετία. Γιατί, γιατί λέει ε, πρέπει να συζητηθεί με τις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν μπορεί να περάσει. Αυτό με το συμπάθειο είναι λάθος είναι μονομερή συμφωνία, είναι μια συμφωνία στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηθεί αυτό το σύστημα και στην περίπτωση που δεν έχουμε τέτοιο σύστημα τότε θα μπορούμε να καταγγέλουμε τη συμφωνία. Και μου είπανε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί η ίδια συμφωνία είναι πενταετής. Και αυτό δεν είναι αλήθεια είναι πενταετής και αυτόματα κάθε χρόνο ανανεώνεται. Δεν έχει λοιπόν δεσμευτική καταληκτική ημερομηνία. Οπότε είναι αδιάφορο αν εμείς ε, θα βάλουμε εκεί 3, 4, 2 ή 7 χρόνια. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μετά μου είπανε ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να καταγγελθεί μόνο ε, με εύλογο λόγο άρθρο 21 άρθρο 21.2 ε, χωρίς κανένα λόγο, με ε, εξάμεινη ε, προθεσμία. Δηλαδή και αυτό ήταν λάθος που μου είπαν ως επιχείρημα. Και από τις 11.30 μέχρι τα μεσάνυχτα που συζητούσα 20 λεπτά στο τηλέφωνο περίπου, ε, μου μπήκανε ψήλοι στα αυτιά ότι δεν την έχουν διαβάσει καν τη συμφωνία αυτή που με παίρνουν τηλέφωνο και θέλουν να φέρουν όχι μένα, το κοινοβούλιο πρώτα τορισμένων γεγονότων. Ότι τώρα ξεκινάει η γραπτή διαδικασία και χάσατε, δεν αλλάζει τίποτα πλέον. Αρκετό καιρό είχαμε την ευκαιρία, γιατί το κοινοβούλιο είναι και πάρα πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ ταχύ στην εργασία του, να το ε, εξετάσουμε. Και όπως ακούστηκε, μπορεί να ακούσετε και από άλλες πολιτικές ομάδες, είχαμε και την πειθαρχία να μην επικρίνουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας, επικεντρωθήκαμε μόνο σε δύο σημαντικά αιτήματα. Το ένα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενδεχομένως ε, ανταποκρίθηκε αλλά δεν έχουμε κείμενο ακόμα για το άρθρο 12 και το άλλο ήταν απέναντι στο Συμβούλιο με τη δεσμευτική ισχύ και την πολιτική πίεση, το μοχλό να μπορούμε να αναστέλουμε ή να καταγγέλουμε τη συμφωνία. Η τριετία έχει πολιτική σημασία, ακριβώς γιατί το ίδιο Κοινοβούλιο το οποίο ζήτησε να αλλάξει η συμφωνία θα είναι το ίδιο το οποίο είναι και υπόλογο και υπεύθυνο να αλλαξει η συμφωνια ειναι το ιδιο το οποιο ειναι και υπολογο και υπευθυνο να ελεγξει ε, αν ε, τα συμφωνηθέντα τηρούνται. Το 2013 λοιπόν θα ήταν αυτό, το ίδιο Κοινοβούλιο, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μεγάλο βαθμό και το ίδιο Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να αναμένουμε από ένα νέο κοινοβούλιο και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξουμε τον ίδιο τρόπο αυτά τα πράγματα. Η όλη τώρα επιχειρηματολογία που λέει ότι ενδεχομένω να καταγγελθεί η συμφωνία κτλ. δείχνει ότι δεν υπάρχει προθυμία στα κρατημέλη να στήσουν ένα σύστημα το οποίο να επεξεργάζεται ε, σε ευρωπαϊκή επικράτεια τα στοιχεία. Για το θέμα της εμπιστοσύνης, πραγματικά πρέπει να σας πω ότι έχει κλονιστεί βαθύτατα. Εχθές είδα τα σχέδια έκθεσης του Κορεπέ και λυπάμαι πάρα πολύ που και η Κομισιόν και η Προεδρία έχουν, την ίδια, έχουν μία διατύπωση προς το Κοινοβούλιο και μία άλλη προς το Συμβούλιο στα έγγραφά τους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι επίπεδο επιτρόπου, σε υψηλότατο επίπεδο, μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα υποβάλει τη θέση ε, του ε, Κοινοβουλίου υπόψη του Συμβουλίου και η Ισπανική Προεδρία δια του πρέσβη είπε ότι θα την υποστηρίξει. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να θεωρώ ότι είναι λάθος ε, τα πλαστά τα έγγραφα αυτά. Ε, βλέπω λοιπόν ότι δεν υποστηρίζεται αυτή η θέση ούτε από την Προεδρία ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά γίνεται συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης γιατί σου λένε είναι αδύνατα αυτά, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ και ξεχάστε τα. Ε, τότε διαρωτώ με γιατί δεν μου το λένε εμένα κατά μούτρα. Τι είναι αυτά τα αδύνατα, έναν ανέφικτο ενδιαφέρουσα ερμηνεία. Πριν από δύο εβδομάδες ότι είναι τώρα πραγματικότητα ήταν επίση ανέφικτο. Το να αλλάξει καν η συνθήκη ή η συμφωνια στο κείμενο. Προχτέ ήρθε ολόκληρο υπάλληλο, τον είπα στην ε, Ένωση για να το αλλάξει αυτό. Και πριν από δύο εβδομάδες πάλι μας λέγατε ότι ήταν ανέφικτη η αλλαγή στο κείμενο του Συμβουλίου. Να όμω που έγινε. Ε, για μένα λοιπόν το ερώτημα. Γιατί αφού έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, να συνεννοούμαστε, γιατί δεν την εκμεταλλευόμαστε, γιατί δεν συζητάμε ε, με εμπιστοσύνη, με ειλικρίνεια και να ανοίγουμε τα χαρτιά μας. Να μην μας διαβεβαιώνετε ότι θα κάνετε το α και μετά πράτε το β. Ξέρετε, θυμίζω ότι είμαστε και στη συναπόφαση και εδώ δεν μπορεί η Προεδρία να ε, υπαγορεύει την ταχύτητα. Θα πρέπει να γίνεται αυτό σε λογική συνεργασία με τα τρία θεσμικά όργανα. Εάν περιμένετε από εμά να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, τότε εγώ περιμένω να μας δώσετε την τρίτη που ζητάμε και επιπλέον και κυρίως το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα είμαι με την πολιτική μου ομάδα στη θαυμάσια πόλη σας Μπιλμπάο για να ψηφίσουμε τον Ιούλιο Κάπως θα πρέπει να αποφασίσουμε εδώ την άλλη εβδομάδα. Ένα ψήφισμα να γράψει κάποιος, ξέρω εγώ. Και εδώ το ανέφεκτο έχει τη δική του ερμηνεία. Είναι εφικτό μέχρι τότε να γράψουμε έκθεση. Πρέπει να μεταφραστεί κιόλα. Και όπως βλέπετε η μετρική μου είναι τα γερμανικά και όχι τα αγγλικά. Άρα θα πρέπει να μεταφράζεται και η έκθεση αυτή. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά. Επιθυμώ να κινηθεί το Συμβούλιο και να μην μας φέρετε ενώπιον και πρώτα τελεσμένων γεγονότων. Και πήρα τηλέφωνο το πρέσβη σας πριν τη συνεδρίαση του Κορεπέρ και όταν έσφιξαν τα πράγματα, σιγεί από το Κορεπέρ. Από τη μία το μεσημέρι προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο τους μόνιμους αντιπροσώπους ε, όταν έμαθα ότι έχει καλώσει η διαπραγμάτευση. Και όταν σε δύσκολου καιρού ε, ε, έχουμε δυσκολίες που μπορούμε εμεί να βοηθήσουμε να λυθούν, περιμένω να σηκώσει ο συνομιλητής μου το τηλέφωνο, το ακουστικό του για να ε, επικοινωνήσει μαζί μου. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώ αξιολογείται τώρα αυτό το πράγμα με ΑΙ. Γιατί αφού είδαμε τι είναι εφικτό και τι είναι ανέφικτο, τα πάντα γίνονται. Ευχαριστώ. Για τους πρασίνους, ο κύριος Ρωμέβα. Sí, Ευχαριστώ πολύ. Έχω καλυφθεί από προλαλήσαντες και μια που δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να επισέλθω κατευθείαν στην ουσία. Κύριε Υπουργέ, για άλλη μια φορά ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ήθελα να σας ε, ε, ξανατονίσω σε συνέχεια να σας είπαμε. Είναι αλήθεια ότι όταν ε, ψηφίσαμε υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα όσον αφορά τα, τις περισσότερες πολιτικές ομάδες όσον αφορά αυτά τα, τις πληροφορίες για τους συμβάτες σε σχέση με το τι ήθελα να μείνει. Διότι αφήσατε το κοινοβούλιο έξω από τη και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν ήταν το μοναδικό, ήταν πολύ σημαντικό, δεν ήταν το μόνο πρόβλημα. Δεν ήταν αυτό η, ο μόνος λόγος που έκανε κάποιες πολιτικές ομάδες όπως εμάς τους πράσινους να εκδηλώσουμε την αντίρρησή μας. Οπότε και τότε είπαμε και τονίσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα ουσίας, το οποίο φοβάμαι ότι ακόμα ισχύει. Δηλαδή ότι ο, τόσο καιρό και τόσους μήνες δεν μας δώσατε κάτι, ένα έγγραφο, ένα ντοκουμέντο, κάτι το οποίο να δικαιολογεί αυτό το οποίο κάνατε. Με αυτόν τον τρόπο που δώσατε τα δεδομένα των επιβατών στις ΕΠΑ. Είπαμε, είναι και θέματα ε, ε δεν είναι τα μόνα. Επομένως, γι' αυτό να δούμε. Να δούμε για ποιο λόγο προβλέπετε να δίνετε τα δεδομένα και να δούμε ακριβώς τι κινδύνους εγκυμονεί αυτό το οποίο κάνατε. Δεν έγινε κουβέντα. Το θέμα δεν επιλύθηκε ακόμα. εκρεμή. Μας τα είπατε κάπως φλού και είπατε ότι τον Ιούλιο πρόκειται να το ξανασυζητήσετε στο Συμβούλιο και φυσικά δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, το είδαμε και θα το ξαναδούμε. Θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε εδώ, στο Κοινοβούλιο, αυτά τα οποία ο κόσμος περιμένει. Άρα χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα και περισσότερη προσοχή. Γιατί εδώ υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Κάτι άλλο τώρα να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο μισό λεπτάκι σε ένα άλλο θέμα. Όσον αφορά τα κέντρα κράτησης ή φιλοξενίας των μεταναστών. Υπάρχουν ε, εκεί κάποια προβλήματα και στην Ισπανία υπάρχουν τέτοια κέντρα κράτησης. Εγώ δεν ξέρω τι έκανε η Προεδρία σχετικά. Πρόκειται να κάνετε κάτι συγκεκριμένο. Προβλέπετε τίποτα για αυτά τα κέντρα κράτηση. Κύριε Κέρχο, έχετε το λόγο. Um, Πρόεδρε, και εγώ με το TFTP θα ασχοληθώ περισσότερο. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις παρατηρήσεις του Υπουργού σχετικά με τις διατλαντικές ε, σχέσεις ε, ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, δηλαδή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διάφορα ζητήματα τρέχοντα που σχετίζονται με την, κατα... την αντιτρομοκρατία, όπου υπάρχει σοβαρή συνεργασία. Θα ήθελα ο υπουργό ε, να σχολιάσει γενικότερα τις συνολικές σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και τη ΣΥΠΑ μετά από την ε, πρόσφατη δήλωση, την πρωτοβουλία PNR για τα δεδομένα της καταστάσης επιβατών και άλλα τρέχοντα ζητήματα. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω στο TFTP. Φυσικά εδώ και καιρό μας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Προφανώς ε, θα συγχαρώ τον συνεισηγητή, τον κύριο Άλβαρο, για τη δουλειά που έχει κάνει. Αν δω τώρα πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν όταν το, το Κοινοβούλιο απέρριψε τις κάποιες προτάσεις, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ με τη ΣΥΠΑ, ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το Κοινοβούλιο, είναι πολύ πιο πρόθυμοι να συζητούν μαζί μας σε σχέση με το παρελθόν. Εντάξει, δεν είχαμε και την ίδια εντολή ε, νωρίτερα. Άλλαξαν τα πράγματα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, τροποποιήθηκαν οι σχέσεις μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τις αρχές ε, τον ΗΠΑ για το χειρισμό της υπόθεσης. Με ανοιχτό τρόπο και διαφάνεια χειρίστηκαν την υπόθεση. Δεν θέλω να σας κατακρίνω, Υπουργέ, αλλά κάποια θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, δυστυχώς δεν μας βοήθησαν τόσο πολύ όσο οι Αμερικανικές αρχές. Αλλά όπως μας υπενθύμησε και ο κύριος Άλβαρο, παρότι πρόκειται για συμφωνία και εγώ είμαι μεταξύ αυτών που πραγματικά πραγματικά ελπίζουν ε, διακαώς ε, να ε, συνάψουμε σύντομα αυτή τη συμφωνία. Είναι μια διατλαντική συμφωνία, αλλά πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα και σε διαθεσμική βάση. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τρόπος χειρισμού αυτών των διεθνών συμφωνιών ποιος πρέπει να είναι. τουλάχιστον στη δική μας ε, πλευρά του Ατλαντικού ε, θα πρέπει να υπάρχει συνένεση και συμφωνία πριν να αρχίσουμε να συζητούμε με τους εταίρους μας ε, στη ΣΥΠΑ. Απογοητεύομαι λοιπόν που πρόσφατα ε, δεν έχουν λάβει υπόψη, έχουν ε, αγνοήσει θα έλεγα κάποιες θέσεις του Κοινοβουλίου. Θα ε, σιωπήσω συνέχεια μετά από κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Θέλω μόνο να πω ότι θα θέλαμε να κλείσει το ζήτημα σύντομα. Ελπίζουμε να κλείσει η συμφωνία τον Ιούλιο γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος. Υπάρχει κενό. Είναι θέμα ασφάλειας. Είναι σοβαρότατο το θέμα. Ε, και δεν πρέπει να υποτιμούμε ε, τα ε, μέχρι τούδε επιτεύγματα μας. Βέβαια, εκκρεμούν ακόμη ένα-δύο ζητήματα που θα θέλαμε να ρυθμιστούν. Κάτι που ήδη αναφέρθηκε, η αναθεώρηση του ζητήματος των τριών ετών. Δεν νομίζω να είναι τόσο ανέφικτο άμα υπάρχει καλή θέληση, αλλά ήδη έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα Παραδείγματο χάρη, η παρουσία της Ένωσης ε, ε, στην ε, άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εάν το χειριστούμε σωστά, εννοώ, θα βελτιωθούν οι σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ και για άλλα ζητήματα, όπου πραγματικά συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της τρομοκρατίας. Γι' αυτό και έχει βαρύτητα το ζήτημα και γι' αυτό πιστεύω ότι ήδη έχει σημειωθεί πρόοδος και θέλω να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να αποτελματωθεί τώρα η υπόθεση. Με λίγη καλή θέληση μπορούμε να τα μεθοδεύσουμε όλα, να τα ρυθμίσουμε όλα πρόσφατα. Ε, έχει οριστεί το χρονοδιάγραμμα, όπως μας είπε ο κύριος Άλβαρο, είναι προς συμφέρον όλων. Όχι μόνο προς συμφέρον της Ισπανικής Προεδρίας, αλλά και προς επερχόμενες Προεδρίες. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες και εδώ και στη ΣΥΠΑ κατά της τρομοκρατίας. Ας μην περιπλέξουμε περαιτέρω το ζήτημα επειδή δεν υπάρχει καλή θέληση. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ταβάρης από την ΚΟΕ τώρα. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για όλες τις ε, διευκρινήσεις σας. Ε, τι γίνεται με την ε, TFTP. Όπως μας είπαν οι Αμερικανοί στην Ουάσιγκτον υπάρχουν 90 εκατομμύρια οικονομικά μηνύματα που αποστέλλονται κάθε μέρα. Χίδιν δεδομένα είναι αυτά, bulk data πάνω από ένα δις μηνύματα το χρόνο. Πάνε στη Λισαβόνα τα μηνύματα, από το Παρίσι πάνε στην, στο Λονδίνο, από το Ντίσελντορφ πάνε στη Βαρσοβία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αυτό δεν αλλάζει. Και αυτό είναι σημαντικό για εδαφικούς λόγους. Θέλουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα να είναι στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και να τα χειριζόμαστε βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό δεν προβλέπεται στη Συμφωνία Πλαίσιο. Θα μας κρίνουν οι πολίτες της Ένωσης από τον Τίσελντορφ, από τη Λισαβόνα, από το Λονδίνο. Δεν ε, θα δίνουν τον κωδικό ε, της κάρτας τους ε, χωρίς να μας κρίνουν. Δηλαδή σας είπα ότι 90 εκατομμύρια μηνύματα περνάνε στη ΣΥΠΑ κάθε μέρα τέτοια οικονομικά μηνύματα. Έχουμε και άλλους σημαντικούς ε, γείτονες, ε, η Ρωσία και εκείνοι έχουν πρόβλημα με την τρομοκρατία και εκείνοι μπορούν να ισχυριστούν ότι απειλούνται από τρίτες χώρες ε, και θα ζητήσουν ακριβώς τα ίδια δεδομένα σε μια ενδεχόμενη συμφωνία και τι θα πει το Συμβούλιο, τι θα... η Ισπανική Προεδρία δεν θα είναι πλέον εκεί, δεν θα έχει πλέον την Προεδρία, τι θα τους πούμε, δηλαδή θα πούμε τα δίνουμε τα δεδομένα στους Αμερικάνους αλλά όχι στους Ρώσους και εκείνοι έχουν δικά τους όπλα για να διαπραγματευτούν. Είδατε ε, πώς χειρίστηκε την υπόθεση του φυσικού αερίου η Ρωσία. Ε, πώς το χειρίστηκε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα. Ε, απομακρύνεται πολύ από τη θέση που θέλουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εσωτερικό το θέμα. Είναι θέμα προστασίας δεδομένων. Και γι' αυτό ανησυχούμε. Και δεν κατοχυρώνεται τίποτα μέσα στη συμφωνία παρά τα ωραία λόγια. Δεν αλλάζει την Αμερικανική νομοθεσία αυτή η συμφωνία. Σε κανένα τη σημείο. Δυνάμει αυτή τη νομοθεσία, ε, οι Ευρωπαίοι που δεν διαμένουν σε Αμερικανικό έδαφο, ε, ε, υφίστανται αυτή την διακριτική μεταχείριση παρά τα ε, περιδικαστικής επανόρθωσης έτσι, που προβλέπονται μέσα στη συμφωνία. Και γιατί λοιπόν η Europol μπορεί να σφραγίζει ε, τα αιτήματα των Αμερικάνων ε, στα πλαίσια του SWIFT. Το να αφήσουμε την Europol να κάνει αυτό είναι σαν να αφήνουμε το μεθυσμένο να φυλάει το μπουκάλι το κρασί η Europol τι θα κάνει, θα πάρει τα μηνύματα που θα στείλουν μετά οι Αμερικάνοι. Μα δεν είναι δικό της καθήκον, δεν προβλέπεται στην εντολή της Europol. Ε, εμείς έχουμε τον Ευρωπα... Ευρωπαίο Επόπτη προστα... Ε, παρακολούθηση και προστασία των ατομικών δεδομένων. Δική του εντολή είναι. Αυτός πρέπει να τα προστατεύσει και το αντίστοιχο Αμερικανικό όργανο. Δεν είναι θέμα της Europol. Ε, τώρα, ποια είναι η εντολή του Συμβουλίου. Ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια αμερόληπτη δικαστική Ευρωπαϊκή Αρχή. Μα το Συμβούλιο πώς αντιλαμβάνεται αυτή την εντολή. Ξαναλέω, δεν είναι δικαστική αρχή η Europol. Παραβιάζεται αυτή η εντολή του Συμβουλίου. Θέλω μια απάντηση γι' αυτό. Η Europol λοιπόν δεν μπορεί να το αναλάβει αυτό. Οπότε τι, τι θα κάνουμε με την Europol. Μα είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Η λισαβονοποίηση της Europol σε αυτό μας οδηγεί. Μα εδώ μιλάμε για συναπόφαση. Ε, μιλάμε για συναπόφαση όμως ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, όχι ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Λευκό Οίκο. Υπάρχουν δύο ζητήματα ε, που ε, ενδεχομένως να ήταν θετικές, αλλά όχι όπως έχουν τώρα. Η παρακολούθηση. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το SWIFT χρησιμοποιείται για τις εμπορικές συναλλαγές. Όπου κι αν είναι, ε, γίνεται η μεταβίβαση των δεδομένων στη Ουάσιγκτον ή οπουδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, εμείς που πήγαμε στην Ουάσιγκτον δεν είδαμε που ακριβώς είναι το κέντρο διαχείρισης των δεδομένων. Μας δείξαν ένα PowerPoint και ένα έντυπο για το αίτημα σε πληροφοριών. Δηλαδή εμά δεν μας έχουν εμπιστοσύνη να μας πάνε στο κέντρο, να δούμε πώς συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Ενώ από πλευρά μα το θέλουν αυτό. Ωραία. Τι γίνεται με το SWIFT. Ε, πρέπει να προσδιορίσουμε τους όρους της παρακολούθησης. Και πώς θα διοριστεί ο υπεύθυνο. Η Επιτροπή θα τον διορίσει. Εάν ναι, θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο. Γιατί θα εκπροσωπεί του Ευρωπαίου πολίτε αυτό το άτομο. Και για να το κάνει αυτό πρέπει να περάσει από το σώμα των αιρετών εκπροσώπων των πολιτών. Αυτό έχει καθοριστική σημασία. Δεν θέλουμε να έρθει κάποιο να μα πει ότι δεν προβλέπεται αυτό. Αυτό δεν είναι υποδιαπραγμάτευση με του Αμερικανού. Χρειάζεται συμβαστική λύση ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό που θα, ε, που θα εκπροσωπήσει του Ευρωπαίου πολίτε στην Αμερική πρέπει να ε, εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, έχει απολύτω δίκαιο ο συνάδελφο Άλβαρο ε, για την ε, προθεσμία που προτείνει. Τρία χρόνια συμφωνία. Αυτό ζητά και έχει δίκαιο. Έχουμε περάσει τόσο καιρό επεξεργαζόμενοι αυτή τη συμφωνία, πρέπει τουλάχιστον να διαρκέσει τρία χρόνια και ξέρετε πόση σημασία έχει αυτό για τα δεδομένα που πρέπει να τα χειριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ε, με θα φύγετε Ωραία. Ε, ε, ε, εσάς σας εκλέξανε για να διοικείτε στην Ισπανία. Άλλο Ισπανία, άλλο Ευρώπη. Εμείς όλοι θέλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβρη, ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να τα θυμούνται αυτά που είπα. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρε. Ο κύριο Μποργέτσιο. Ευχαριστώ Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα μακρηγορήσω. Ο ισπανικός λαός μου είναι πάρα πολύ προσφυλής και αγαπητός. Και θα θέλαμε να απευθύνουμε και τα συλληπιτήριά μας για το δυστύχημα που έγινε σήμερα. Και θα θέλαμε να σας καλέσουμε να εγκρίνετε ε, πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας ε, για ε, τους σιδηροδρόμους και ιδιαίτερα τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Για τη λαθρομετανάστευση στη Μεσόγειο, όταν έγινε απόπειρα να σταματήσει η σκανδαλώδης αυτή η κατάσταση με την εμπορία ανθρώπων, οι συμφωνίες που συνήφθησαν ήτανε ο Ιταλός Υπουργό Μπαρόνι και η Ιταλική κυβέρνηση έχουν συνάψει πολύ σημαντικές συμφωνίες με τη Λιβύη. Και τελικά σταμάτησαν να έρχονται πλοία με ε, λαθρομετανάστες. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτή τη στρατηγική. Δεν νομίζετε ότι τα κράτη που αντιμετωπίζουν αυτή την εγκατεπίγουσα κατάσταση και την πίεση, η Μάλτα, η Ιταλία, η Ελλάδα, δεν αξίζουν ε, καλύτερη υποστήριξη και μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πού είναι η περίφημη ευρωπαϊκή στρατηγική ε, απέναντι σε αυτά. Πού είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μάλλον, πολύ αργή είναι η πρόοδος. Τα αποτελέσματα που έχουν τα κράτη-μέλη, αν υπήρχε όντως ευρωπαϊκή στρατηγική, θα ήταν πολύ καλύτερα. Να δούμε και ποιες είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής, χώρας με τις τρίτες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες και χώρες διέλευσης. Τις βοηθάμε οικονομικά. Είναι υποδειγματικές οι Ιταλικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, το ξαναλέω. Θα ήθελα επίσης κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο για το σλόγγαν που ε, αναφέρατε προηγουμένως. Πυγμή και ανεκτικότητα απέναντι στη θερμοκρατία. Δεν έχουμε δικτατορίες στην Ευρώπη, δεν έχουμε καραπίνο σετ. Η ανεκτικότητα, η ανοχή είναι κάτι το δεδομένο, δεν χρειάζεται να το εξαγγέλουμε. Όταν όμως είναι τόσο μεγάλη η ε, απειλή όσο από την τρομοκρατία θα πρέπει όντως να επιδεικνύουμε πυγμή. Γιατί δεν θέλω εγώ υπό το μανδύα της ανοχής και της ανεκτικότητας να... να θεωρούμε ότι τα Ισλαμικά κέντρα, τα τεμένη είναι κάτι το ιερό που δεν μπορεί κανείς να θίξει, να πειράξει να έχουμε τέτοιες ε, ζώνες άσυλα τρομοκρατίας. Είτε πρόκειται για τη βασική τρομοκρατία, την ισλαμική τρομοκρατία, από όπου και αν προέρχεται. Και για να επανέλθω στο SWIFT και στο TFTP, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υπογράψει αυτή τη συμφωνία, να επιδείξει πυγμή και σθένος, είναι πρόοδος και η διεθνής εγκληματικότητα πάρα πολύ επικίνδυνη. Ας σκεφτούμε και τους μελλοντικούς κινδύνους. Κινδύνους τρομοκρατικών ε, ε, ενεργειών με χημικά και άλλες επικίνδυνες ουσίες. Ας προχωρήσουμε λοιπόν προς τα εμπρός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόγκς από τους μη εγγεγραμμένους.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 freedom of expression. Διευκολύνουν αυτές οι αξίες που είπατε την ελευθερία του συναθρίζεστε και ε, άλλες δημοκρατικές αξίες και από την άλλη τις ουσιαστικές αξίες, όχι τις διαδικαστικές, δηλαδή αυτές που είναι πιο ουσιαστικές για τη λειτουργία της δημοκρατίας και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε σαν ο κοινωνικός φιλελευθερισμός είναι αυτές οι αξίες που πάρα πολλοί τις τιμούν, αλλά τελικά ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι αυταπόδεικτες. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι υπάρχει συνένεση για αυτές τις αξίες αυτό είναι η συνταγή ούτως ώστε τα κοινοβούλια να γίνονται Σοβιέτ κεντροκατευθυνόμενα όπως και να όπως και να το δικαιολογεί και αυτός επομένως αυτές οι διαδικαστικές δημοκρατικές αξίες να θεωρήσουμε ότι είναι αυταπόδεικτες ότι όμως παρόλα αυτά δεν θα πρέπει κανείς να περιορίζει την συζήτηση επιβάλλοντας κάποιες ε, αξίες, κάποια δίκτυα, κάποιες ιδέες, κάποιες, ε, ε, κάποιες προκαταλήψεις που σταματούν τη συζήτηση, το διάλογο και άρα το να οδηγεί κανείς σε αναγκαστική επιβολή κάποιες κοινωνικής πολιτικής μπορεί να οδηγήσει ε, όπως το είδαμε σε πολλές χώρες μέλη, το να χτυπιέται ο συνδικαλισμός και τα σχετικά δικαιώματα. Δεν λέω ότι κανείς εδώ είναι κακόπιστος. Νομίζω ότι όλοι ξεκινούν με τις καλύτερε προθέσεις του έργου τους, όπως η και Προεδρία. Όμως, θα πρέπει για τα θεσμικά όργανα να θεωρήσει κανείς ότι βάση κάθε ενέργειας είναι μια ατζέντα, μια μέση διάταξη που διαπνείται από φιλελεύθερο πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και τώρα για αυτό τον πρώτο γύρο τραπέζι θα λάβει το λόγο ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χωρίσω τις απαντήσεις μου σε δύο μέρη. Σε δύο μέρη Πρώτα πρώτα να σας πω για τους εκπροσώπους των κομμάτων που αναφέρθηκαν σε αυτά τα οποία είπα εγώ στην εισηγησή μου. Στη συνέχεια να απαντήσω στους άλλους που αναφέρθηκαν στο SWIFT. Μιλήσατε για το SWIFT μερικοί από εσά στις ερωτήσεις που υποβάλατε πρώτα πρώτα να πω για τον κύριο Ντία Ντεμέρα ότι τον ευχαριστώ πρώτα πρώτα διότι γενικώ συμφώνησε με τα όσα έκανε η Ισπανική Προεδρία. υπέβαλε κάποιες παρατηρήσεις, ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις και ξεκίνησε με το θέμα του ασύλου. Δηλαδή για το ότι η Ισπανική Προεδρία πρόθεσε την υλοποίηση αυτού του Ευρωπαϊκού Συστήματο χορηγή του Ασύλου μέχρι το 2012. Κάποια πράγματα που διεκπαιρεώσαν που τα είχε αφήσει εκκρεμή η, η Σουηδική Προεδρία και όπω το είπαμε κατά την Προεδρία, πρόκειται για περίπλοκο θέμα. Το άσυλο είναι δύσκολο. Λεπτό. Έχουμε διαφορετικές ευαισθησίες από πλευράς κάθε χώρα και αυτό μας οδηγεί πολλές φορές σε σύγκρουση και ανταγωνισμό. Άλλα προσβεύει η Προεδρία, άλλα η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη, άλλα. Γι' αυτό σας λέω το θέμα είναι περίπλοκο. Τι κάναμε εμείς όμως. Εμείς επιλύσαμε κάποια προβλήματα, κάποια τα οποία ήταν όριμα προς επίλυση, όπως ας πούμε αυτή η υπηρεσία της Μάλτας για την πλαισίωση και υποστήριξη. θα είμαστε στην φάση ορισμού και διορισμού του εκεί επικεφαλής και αυτό θα διευκολύνει θεωρούμε την συνεργασία των ε, χώρων επίσης είπαμε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την εμπειρία μας και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αντιστοιχεί σαν πρικοδότηση σε αυτό το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δεν το είπατε, αλλά απορρέει από αυτά τα οποία είπαμε. Τώρα έχουμε κάποια άλλα θέματα τα οποία εκκρεμούν, τα οποία όπως και ο ίδιος προανέφερε είναι διάφορα. Έχουμε δύο κανονισμούς και τρεις οδηγίες. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι μέσα από τα νομοθετήματα που έχουμε και με τους κανονισμούς και με τις οδηγίες κάτι να βγει. Οπότε, μέσα από την ομάδα εργασίας για το άσυλο, αλλά και την Στρατηγική Επιτροπή, προσπαθήσαμε μια σειρά συναντήσεων, με τη βάση ενός χρονοδιάγραμματος, να προχωρήσουμε. Δεκάδες ήταν οι συναντήσεις που έγιναν και με το Ομάδα και αυτήν και με την Στρατηγική Επιτροπή. Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε ενενετικές θέσεις. Έχουμε τώρα δύο οδηγίε που προωθήθηκαν γιατί θεωρήσαμε ότι είχαν κολλήσει όσον αφορά την υποδοχή των μεταναστών και των ετούντων άσυλο. Θέλουμε να υπάρχει όσο γίνεται πιο ομοιογενής προσέγγιση όπως είπε και ο κύριος Μωράες. Αυτό προσπάθησε να κάνει η Ισπανική Προεδρία. Η δέσμη όλων των μέτρων για το άσυλο προσπαθήσαμε να προχωρήσει με τρόπο ομοιογενή. Γι' αυτό δεν θα αφήσουμε τη μία οδηγία για να προωθήσουμε την άλλη. Ταυτόχρονα επομένω, εξετάσαμε και τις τρεις οδηγίες. Τι έκανε επομένως η Προεδρία. προσπαθήσαμε να είναι στην ίδια φάση εξέλιξης αυτές οι δύο οδηγίες, όπως και η οδηγία για την υποδοχή, που ήταν αυτή που είχε ξεκινήσει και είχε προχωρήσει περισσότερο. Το ίδιο αφορά και στον κανονισμό του Δουβλίνου. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ισχύει. Δεν σας κρύβω ότι ακόμα υπάρχουν διαφωνίες για ουσιαστικά θέματα. Οριζόντια θέματα αφορούν όλες αυτές τις οδηγίες για το κοινό σύστημα του ασύλου, όπως ας πούμε τι ορίζεται μέλος οικογενείας. Είναι κάτι που και τα κρατημέλη, δηλαδή το με τι προϋποθέσεις, με τι εγγύσεις χορηγείται το άσυλο. Τι γίνεται όσον αφορά την αναστολή ισχύω του κανονισμού του Δουβλίνου όταν κάποια χώρα το ζητήσει για τους προβλεπόμενους λόγους. Άρα προωθήθηκαν στον ίδιο βαθμό όλες αυτές οι οδηγίες για το άσυλο. Με τίποτα δεν είναι εύκολο το έργο μας, όμως όπως προείπα. Δεν αναφέρθηκε το ο συνοδευτούς ανηλίκους γιατί μίλησε γι' αυτό εχθές η συνάδελφος που ήρθε να σας δει για την αστυνομική συνεργασία μου, πια ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ομάδων έρευνας και ομάδων ε, συνεργασίας, γιατί εδώ έχουμε και το θέμα της συνεργασίας αστυνομικών με δικαστικούς. Αυτό είναι οι ομάδες έρευνας, ενώ η, συνεργασία των αστυνομικών είναι η συνεργασία αστυνομικών με αστυνομικούς. Να, ας πούμε, σαν παράδειγμα, έχουμε ε, κάποια συμβάντα τα οποία λαμβάνουν χώρα σε ένα ε, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είχε γίνει για το κύπελο εθνών στην ε, Αυστρία. Εκεί είχαμε συνεργασία των αστυνομικών. Ενώ αντίθετα, ας πούμε για να κατοπολεμήσουν την ΕΤΑ, έχουν συνεργαστεί με τους δικαστέ και με τους αστυνομικού, οι Ισπανοί με τους Γάλλους. Δηλαδή, Στη μία περίπτωση έχουμε ερευνητικέ ενέργειε, στην άλλη έχουμε κάποιε ενέργειε καταστολή των διοικητικών αρχών, όπω είπαμε σε κάποιε διοργανώσει, ε, όπου αυτό το οποίο εξυπηρετεί είναι να έχουμε αστυνομικού από όλε τι εμπλεκόμενε χώρε. Γιατί ακριβώ εκεί υπάρχουν ε, άνθρωποι από περισσότερε χώρε. Όσο αφορά τώρα το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, εδώ νομίζω ότι προχωρήσαμε πολύ. Επίσης ε, όσον αφορά το, μαύρο χρήμα, έχουμε κάνει και εδώ πολλά. Μας απασχόλησε και βέβαια όπως είναι λογικό συνεργαστήκαμε με ε, αστυνομία πολλών χωρών μελών. Και εδώ είχαμε κάποιες ε, πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις με επιτυχία. Για τη Europol. Είπαμε ότι μέχρι το 2013 θα έχουμε τον νέο κανονισμό. Αν με ρωτάτε βεβαίως, όπως ε, ε, ήταν η θέση μας ανέκαθεν, θέλουμε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές της. Ευχαριστώ τον Κλοντ Μωράς για τα καλά του λόγια όσον αφορά το έργο που επιτελεί η Προεδρία. Όντως, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης τα καλύπτει όλα. Εκεί καλύπτονται όλα όσα θέλουν τα κράτη-μέλη. Να ένας τρόπος να πετύχει κανείς ομοφωνία. Βέβαια ένα πρόγραμμα δράσης πρέπει να έχει κάποιες προτεραιότητες. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό έγινε με το σωστό τρόπο. Έχουμε προτεραιότητες, έχουμε και χρονοδιάγραμμα, έχουμε ανάληψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων, επομένως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό κείμενο ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό το γενικό πρόγραμμα θα λάβει σάρκα και ωστά από όλες τις ιδιωτικές αρχές, τις αρχές που φροντίζουν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. νομοθεσία το τι γίνεται με την οργάνωση των Υπουργείων. Ξέρετε, το κάθε, η κάθε χώρα, κάθε κράτο μέλος έχει άλλη οργάνωση όσον αφορά τα Υπουργεία της. Ε, ας πούμε στην Ισπανία ο κανόνας είναι να έχουμε χωριστό Υπουργείο Ιστορικών και χωριστό δικαιοσύνη. Αλλού όμως ισχύει το αντίθετο. Άρα αυτή η κατάσταση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μεσοπρόθεσμα εγώ θεωρώ ότι πιο πολλά είναι τα υπέρ παρά τα κατά. όμω είναι αλήθεια ότι πρόθεσμα το να γίνεται ένας χωρισμός αυτών που πριν δούλευαν από κοινού αυτό λογικά μας πήγε πίσω. για τη δέσμη για το άσυλο, σας είπα τη γνώμη μου, αλλά κάποια στιγμή πάντω θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να θεσπιστεί μια οδηγία, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όταν έρθει η ώρα να έχουμε όλα τα κοινά στοιχεία, ε, όταν έχουμε και τις τρεις ε, οδηγίε έτοιμε να κάνουμε αναθεώρηση των συμφωνιών, να δούμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία, ποια είναι τα, τα οριζόντια θέματα και όταν τα έχουμε κλείσει τότε είναι λογικό ότι πρόκειται να περάσουν αυτές οι οδηγίες. Και τέλος, ρώτησε κάποιος κάτι. Ε, έγινε μια αναφορά από τον κύριο Ρωμέβα για τα κέντρα προσφύγων δεν ξέρω πώς ε, λειτουργούν σε διάφορα κράτη-μέλη Ξέρω ότι γίνεται στην Ισπανία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με τον Ερυθρό ε, Σταυρό. Ε, δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κατάσταση σε άλλες χώρες. Ε, οι επόμενες παρεμβάσεις ήταν ε, για το SWIFT. Μα αυτά τα έχει συζητήσει με την κυρία Μάλστρον και ε, στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να πω δύο-τρία στοιχεία μόνο και να κάνω και κάποια αναφορά στην τελική τοποθέτηση του κυρίου Άλβαρο, γιατί αυτή δείχνει τις δυσκολίε που υπάρχουν αυτό τον καιρό να προχωρήσουμε. Πρώτον, η αλήθεια είναι ότι βιαζόμαστε. Δεν βιάζεται η Ισπανική Προεδρία, που βιάζεται και αυτή βέβαια, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες αδειμονούν στα κράτη-μέλη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί είναι γεγονό ότι ένα εργαλείο σαν το TFTP ε, βελτίωση τη ασφάλεια, γιατί το πιστεύω ότι τη βελτιώνει, ε, μα χρειάζεται και αυτή τη στιγμή είναι ε, διακεκομένο. Έχει σταματήσει η λειτουργία από το Φεβρουάριο, δεν διαβιβάζονται τα στοιχεία και είναι λιγότερη ασφάλεια, μου επιτρέπετε. Σχετική ασφάλεια είναι τώρα σε σχέση με το Φεβρουάριο. Βιαζόμαστε, βιαζόμαστε. Και η Ισπανική Προεδρία. Είναι θέμα ευθύνη όμω αυτό όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, χρειάζεται επιτάχυση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι το ξέραμε, γι' αυτό έχουμε εργαστεί όλοι πάρα πολύ γρήγορα. Και αν δει κανεί τα ενδιάμεσα ορόσημα που είχαμε βάλει για ευρωπαϊκή ε, λειτουργία, αυτό είναι πραγματικά τροχάδι. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή στις 10 Μαΐου, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρόταση της 24 Μαρτίου, 10 Μαΐου το Συμβούλιο το ενέκρινε, 8 Μαΐου το Κοινοβούλιο είχε γκρίνει ψήφισμα για την εντολή, είμαστε Ιούνιο και μιλάμε ήδη για συμφωνία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά κατεπίγουσα η διαδικασία και θα πρέπει επιγόντως να αντιδράσουμε, γι' αυτό ε, και το πράττουμε γρήγορα με ευθύνη και από τούτη την πλευρά του Ατλαντικού αλλά και από την άλλη. Στη συνέχεια, άλλο γενικό θέμα. Άλλαξε το προσχέδιο της συνθήκης που έχουμε αυτό το καιρό και που το κοινοβούλιο απέριψε. Άλλαξε, άλλαξε ουσιαστικά προς την κατεύθυνση που ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί το Κοινοβούλιο πέριψε τη συμφωνία. Η Κομισιόν είχε πει ναι. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όχι. Λοιπόν, οι αλλαγές που μπήκαν στη νέα συμφωνία είναι καρπός των ε, όσων ζήτησε το Κοινοβούλιο και της άρνησης του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει και δημόσια αυτό να το ανακοινώνουμε. Άλλωστε, μεταξύ αυτών απερίφθηκε δική μου πρόταση υπουργική και δεν έχω κανένα πρόβλημα το να γνωρίζω. Βεβαίως υπήρξαν σημαντικές αλλαγές και έμεσα αναγνωρίζεται η αρχή της ε, αναλογικότητας που δεν υπήρχε, μεγαλύτερη διαφάνεια της εποπτείας της ΗΠΑ γιατί το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον θα παρεμβαίνει και αυτή και να υπάρχει ένα TFTP ε, ευρωπαϊκό που θέλουμε όλοι να γίνει ε, σημαντικές βελτιώσεις στην προστασία των δεδομένων ε, σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς που έχουν τη διοικητική και δικαστική επίβλεψη Όλα αυτά είναι στοιχεία πραγματικά πρόοδου. Υπάρχουν και ε, αντικειμενικοί περιορισμοί για διαβίβαση στοιχείων σε τρίτες χώρες. Πολλές λοιπόν από τις προφυλάξεις και τις ασφαλιστικές δικλίδες που θέλαμε μπήκανε για την πεταετία αυτή. Συνοψίζω, είναι διαφορετική η συμφωνία αυτή τη FTP από την αρχική, την οποία το κοινοβούλιο σας απέρριψε. Είναι πάρα πολύ διαφορετική. Και εδώ έχουμε πολλά στοιχεία του κοινοβολίου, πολλές προβλέψεις του Κοινοβουλίου, διότι το Το θέμα της διαπραγμάτευσης έγινε πολύ καλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένε Πολιτείε επέδειξαν ευελιξία. Θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Η κυρία Μάστρομ ήρθε εδώ, δεν απατώμε, στις 9 του μηνό Ιουνίου και εξέθεσε τις βασικές γραμμές συμφωνίας που τότε δεν είχε υπογραφεί ακόμα, έδειξε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 10 του μηνός ε, συνεδρίασε με τις πολιτικές ομάδες και ξέρω ότι η συμφωνία που είχε γίνει άλλαξε, σα είπα, ακριβώ, βάσει των όσων ζητήσατε εσείς και από την κυρία Μάστρομ. Και το Συμβούλιο επίσης ήθελε να, να είναι αντανάκλαση και των πολιτικών ομάδων ενσυχίε και των όσων θέλουν τα κράτη-μέλη. Και κάναμε λοιπόν αλλαγέ και από το Συμβούλιο ακριβώ για να ικανοποιήσουμε τι κοινοβουλευτικέ ομάδε που ακόμα δεν είχαν συμπεριληφθεί τα ε, λήματά του και τα αιτήματά του στο κείμενο. Έχει δίκιο ο κύριο Άλβαρο όταν λέει ότι πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι Ηνωμένε Πολιτείε και τώρα θα πρέπει να ξανανοίξει η συζήτηση και η συμφωνία και ξανά ανοίξε. και άλλαξε και το άρθρο 12 εδάφιο 1 για να καταλάβουμε ότι κάποιο που θα εκπροσωπεί την, Κομισιό, μάλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση διορθώνει ο Υπουργό, θα ε, είναι στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, την ώρα που θα χειρίζονται και θα επεξεργάζονται μαζί με την εταιρεία SWIFT τα στοιχεία. Δηλαδή κάποιος εντεταλμένος Ευρωπαίος καθημερινά θα είναι στις ΗΠΑ και θα επεξεργάζει τα στοιχεία. Και αυτό ακριβώ ανταποκρίνεται στις προτάσεις του Κοινοβουλίου που άλλαξε αυτή τη στιγμή ήδη είχε υπογραφεί η συμφωνία και καταφέραμε να πείσουμε και τις ΗΠΑ να ξανανοίξει και να αλλάξει συμφωνία. Και είναι γεγονό ότι το Συμβούλιο προσπάθησε να βάλει και κάποια άλλα πράγματα που ζητούσαν οι πολιτικές ομάδες. Γι' αυτό κάναμε με όλες τις πολιτικές ομάδες ε, επαφές και με τον κύριο Άλβαρο εγώ επανειλημμένα είχα συζητήσει. Βάλαμε ας πούμε δήλωση συμφωνίας του Συμβουλίου έτσι ώστε αν κάποια μέρα έχουμε συνολική μεταφορά των στοιχείων στις ΗΠΑ αυτό να ε, περιλαμβάνεται στη συμφωνία και να προβλέπεται. Και το μέλημα αυτό του Κοινοβουλίου το έχουμε βάλει. Ε, υιοθετεί το Συμβούλιο λοιπόν αυτή την ανησυχία και είναι πάρα πολύ λογικό. Εάν έχουμε συνολική συμφωνία με τους Αμερικανούς για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει αυτό να φαίνεται και στη συμφωνία. Το είπαμε άλλωστε. Γι' αυτό μπαίνει Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή ανησύχησε το Κοινοβούλιο. Για την Ευρωπόλ επίσης ακούστηκαν διάφορα ανησυχίε. Ξέρετε ότι έχει δικαστικό έλεγχο, το θυμίζω σε κάποιο βουλευτή που αναφέρθηκε. Η ε, ε Ευρωπόλ έχει βεβαίω δικαστικό έλεγχο. Ό,τι κάνει υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Αλλά είναι γεγονό ότι κάποιοι ανησύχησαν για το ρόλο τη Ευρωπόλ. Και είναι και πάλι κοινοβουλευτική ανησυχία, αλλά και από κάποια κράτη-μέλη. Γι' αυτό εγκρίναμε και μια άλλη απόφαση στο Συμβούλιο, όπου σαφώς ορίζεται με ποιο τρόπο λειτουργεί η Ευρωπόλ και γιατί θα ελέγχει η Ευρωπόλ αυτά που ζητάν τα κράτη-μέλη και κατά πόσο προσαρμόζονται στη συνθήκη. Προσοχή, σας θυμίζω ότι δεν μπαίνει στην ουσία η Ευρωπόλ προς το παρόν, ελέγχει το τυπικό σκέλος. Έτσι, εάν οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, συμμορφώνονται με τα όσα έχουμε συμφωνήσει και υπογράψει μαζί τους. Έτσι λοιπόν, δύο είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου που προσπάθησαν την τελευταία εβδομάδα να ε, λάβουν υπόψη τους τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και τροποποιήθηκε το άρθρο 12 για να ε, μπει αυτή η βαθύτατη ανησυχία του Κοινοβουλίου για τον έλεγχο των δράσεων και των συναλλαγών SWIFT στι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπήρξαν κάποιε προτάσει, είναι γεγονό του κυρίου Άλβαρο και το συζητήσαμε μαζί του. Πρέπει να σα πω ότι το Συμβούλιο έτεινε βίκό ου στα όσα ζήτησε. Ναι, κύριε Άλβαρο, ναι. Σα το λέω. Μην αντιδράτε, το κάναμε. Τώρα 100% δεν τα υιοθετήσαμε αυτά που ζητάτε, αλλά μερικά από αυτά που ζητάτε τα ακολουθούμε. Παράδειγμα, βάλαμε στην απόφαση του Συμβουλίου, στην απόφαση του Συμβουλίου, στο δεύτερο άρθρο, υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του χρόνου να φέρει ένα νομικό ε, δικαστικό σύστημα για να, ε, ένα νομικό σύστημα για το πώς θα μπει ε, και στην Ευρώπη αυτό το TFTP. Είναι απόφαση δεσμευτική, την πήραμε χτες, συζητώντας με τον κύριο Άλβαρο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνοψίζω, αυτό που φάνηκε ως συμπέρασμα του Συμβουλίου και απλή σύσταση μετά τη χθεσινή απόφαση του Κορεπέρ είναι άρθρο. Έχει μπει στο διατακτικό. Είναι νομικά δεσμευτικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι ώστε θα πρέπει να βάλει το νομικό πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή TFTP που είναι το πρώτο αναπόφευκτο βήμα έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να υπάρξει στην Ευρώπη. TFTP. Και έχει ένα χρόνο στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάζουμε και προθεσμίες. Τις λέμε σε ένα χρόνο θα πρέπει να μας έχει φέρει σε όλα τα θεσμικά όργανα αυτό το πλαίσιο για να μπορεί να εφαρμοστεί η TFTP στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, βάλαμε και ένα τρίτο άρθρο στην απόφαση και αυτό το τρίτο άρθρο τι λέει, ότι αν σε πέντε χρόνια που τόσα ε, ισχύει η συνθήκη δεν υπάρξει ευρωπαϊκή TFTP να ληφθεί υπόψη. Μάλλον όχι. Όταν έχει συσταθεί αυτή η ευρωπαϊκή TFTP θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στη συμφωνία με τους Αμερικανούς και μπορεί να αναθεωρηθούν ορισμένα, ας πούμε ο ρόλος της Ευρωπόλ σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, το στοιχείο που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γιατί πενταετία, διότι πέντε έτη είναι η διάρκεια τη συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι γεγονό ότι μπορεί να αναθεωρηθεί. Μπορεί, δεν αμφιβάλλω, κάθε έξι μήνε σύμφωνα με την ίδια τη συνθήκη. Αλλά αυτό που δεν μου φαίνεται λογικό και θέλω να το πω με κάθε σαφήνεια στο Κοινοβούλιο είναι να πάρουμε νομικά δεσμευτική απόφαση που βασικά θα λέει το εξής. Εάν η Ευρώπη δεν οργανώσει το FTP το ευρωπαϊκό, σε τρία χρόνια ε, να στέλνουμε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τι λέμε, όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τη συμφωνία στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα είναι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πενταετούς διάρκειας να διαρκεί τρία χρόνια. Ε, αυτό πηγαίνετε να το εξηγήσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά δύσκολο. Είναι ένα είδος μονομενούς αναθεώρησης ε, από μια πενταετία στην τριετία. Αναθεώρηση βάσει των όσων θα κάνουμε εμείς οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Και εάν αδρανήσουμε υποχρεωτικά δηλαδή θα αναθεωρήσουμε μια πενταετή συμφωνία πάνω στην τριετία. Αυτό δεν μπορούμε να το υπερασπιστούμε απέναντι στους Αμερικανούς. Και θέλω να σας πω επίσης ότι η τριετία ποτέ δεν εμφανίστηκα ε, και παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες της διαπραγμάτευσης. Πουθενά δεν έλεγε η ευρωπαϊκή απόφαση ε, του Κοινοβουλίου, ούτε η αρχή που έκανε τη μελέτη. Μιλάει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ε, ποιο είναι το εύλογο. Η τριετία είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Και Νομίζω ότι δεν έχει λόγο ύπαρξη. Δεν θα μπω στη νομική συζήτηση, θα μπορούσα να την κάνω. Γιατί ορισμένοι νομικοί του Συμβουλίου λέγουν ότι και αυτή η διατύπωση όπως προτείνεται δεν ευσταθεί, διότι είναι αντιφατικό με τη διάρκεια της ίδιας συμφωνίας. Δεν μπαίνω, λέω, σε αυτή τη νομική συζήτηση που θα ήταν συναρπαστική από πλευράς νομικής, αλλά από πλευράς πολιτικής είναι μια ρήτρα αναθεώρησης μονομερής συνθήκη συμφωνίας πενταετούς διάρκειας με τις ΗΠΑ και εμείς τη λέμε ξαφνικά μετά από τρία χρόνια την αναθεωρούμε αν δεν κάνουμε ευρωπαϊκή TFTP. Κατανοείτε ότι είναι αρκετά περίπλοκο αυτό να το υπερασπιστούμε απέναντι στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή μετά από μήνες συζητήσεων. Και αφού έχουμε υπογράψει πενταετή διάρκεια τη συμφωνίας. Φανταστείτε επίση, κυρίε και κύριοι, ότι θα υπήρχε η δυνατότητα. Τελειώνω, πρόεδρε, ναι, ναι, τελειώνω. Θα υπήρχε δυνατότητα, λέγω, ε, εάν κάποιο από τα ευρωπαϊκά κράτη ήθελε να διαρκέσει μόνο τρία χρόνια η συμφωνία με την Αμερική, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή TFTP. Αρκεί ένα θεσμικό όργανο ή κάποια κράτη-μέλη να επιθυμούν τριετία αντί για πενταετία, αρκεί να μπλοκάρουν ε, τη δημιουργία της TFTP της Ευρωπαϊκής για να το πετύχουν. Δηλαδή, δίνουμε στην Ευρώπη πλέον τη δυνατότητα να εξαντλήσει ε, αυτή τη στάση της. Ε, έχουμε υπογράψει συμφωνία για πέντε χρόνια, δεν μπορούμε να τρέψουμε στα τρία ε, έτη. Και σας λέω ότι αυτό μας προέκυψε τελευταία στιγμή. Έγινε αναθεώρηση του άρθρου 12.1. Λήφθησαν υπόψη τα μελήματα ε, του Κοινοβουλίου. Ε, συμμετέχει η Ευρωπόλ. Νομίζω ότι πλέον η συμφωνία είναι καλή και περιλαμβάνει ε, τα όσα θέλουμε. Καμιά συμφωνία και καμιά συνθήκη δεν ικανοποιεί 100% όλα τα μέρη, αλλά έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια και αξίζει πραγματικά τον κόπο να εγκρίνουμε τη συμφωνία που σε μεγάλο βαθμό, όχι ε, βέβαια 100% έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ και αλλού. Ευχαριστώ για την επική σας πρόεδρε. Κυρίες και ο πρόεδρος, ε, πάμε πάρα πολύ χάλια από χρόνο. Ε, είμαι βέβαιος ότι όποιος του περιορίσουμε το χρόνο αγόρευσης θα εκφράσει παράπονα ότι δεν μπορεί να εκφραστεί για ένα θέμα που είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ επίμαχο. Από τα πιο επίμαχα που έχουμε συζητήσει τον περασμένο χρόνο στο Κοινοβούλιο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι ανεξάντλητος. Κλείνει ο κατάλογος για δεύτερο γύρο και θα σας κόβω στο δίλεπτο για να μπορέσει στη συνέχεια να απαντήσει ο υπουργό. Θυμίζω ότι αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει επανειλημμένα πάρα πολλές φορές. Έχουν ακουστεί όλες οι απόψεις, σίγουρα δεν πρόκειται να ακούσουμε τίποτα καινούριο. Θα είναι πάντα επανάληψη παλαιότερων τοποθετήσεων σε ε, διάφορα επεισόδια του σύριαλ αυτού της συζήτησης για το θέμα, το τόσο ευαίσθητο. Λοιπόν, να, κοιτάξτε, κοιτάξτε, κύριε Ταβάρη, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, το θέμα το έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά, δεν είναι πρώτη φορά. Μα έχουμε δώσει επανειλημμένα το λόγο. Αφήστε με να θέσω ένα διαδικαστικό. Μα ε, υποσχεθήκατε στη μέση διάταξη να έχουμε ένα σημείο για το TFTP. Ήταν στη μέση διάταξη χτε τη Επιτροπή μα. Αναβλήθηκε για σήμερα και τώρα εξαφανίστηκε το σημείο του TFTP. Έτσι, ο Υπουργό μπορεί να μην απαντήσει για τη λισαβονοποίηση του ρόλου τη ε, Europol. Μα είναι κέρια σημασία. Σα παρακαλώ, θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά ότι πρέπει να ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία γνωμοδότηση για την ε, λισαβονοποίηση, για τι αλλαγέ στην εντολή τη Europol ε, μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πρόεδρο, ναι, ναι, ένα λεπτάκι και θα σα πω. Ε, ο κύριο Αλβαρό κανονικά είχε ανηλυμένη υποχρέωση στι 9, τέλο πάντων ήρθε στι 9 και 4. Αλλάξαμε τη σειρά συζήτηση και ε, εισαγάγαμε το TFTP στη συζήτηση και τώρα θα κάνουμε γενική συζήτηση, όχι μόνο για τα συμπεράσματα και τα αποτέλεσμα της Ισπανικής Προεδρίας αλλά ε, ε, και για το TFTP. Σας παρακαλώ δύο λεπτά χρόνος αγόρευσης κατανότατο όριο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπουζουτήλ, ευχαριστώ ε, τον ε, Υπουργό. Ε, εκτιμούμε τις προσπάθειες που κάνατε, κυρίως για το SWIFT και τις προσπάθειες που έκανε η Προεδρία τις τελευταίες ημέρες. Αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Τζόναθαν Φόλ για τη δουλειά που έχει κάνει σε αυτό το θέμα, αλλά και γενικότερα στην Γενική Διεύθυνση ΔΕΗ. Θα μας λείψει ε, στην Επιτροπή και ε, κάποια μέλη μπορεί να τρέξουν από πίσω σας στην ΙΜΚΟ, να σας τυχιώσουν. Ε, λοιπόν, θα περιοριστώ στο θέμα FTP. Συμφωνώ με σας, Υπουργέ, ότι σημειώθηκε βασική πρόοδος, ένα σημαντικότατο επίταυμα και έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ από το Φεβρουάριο. Επειδή τώρα είμαστε στα πρόθυρα της διετής προσέγγισης, αυτό δηλαδή που επιθυμούσε το Κοινοβούλιο, αφ, δεν θα ήταν μεγάλη νίκη για μας. Τι εννοώ με αυτή τη, διαδικασία. Αφενός ε, επιτρέπουμε την μεταφορά των χίλιων δεδομένων, αλλά υπό δύο όρους, ότι η μεταφορά θα γίνεται υπό αυστηρότητα τους ελέγχους και δεύτερον αναλαμβάνουμε ε, την δέσμευση να διακόψουμε αυτή τη μεταφορά χίλιων δεδομένων όταν θα αρχίσει να υλοποιείται η TFTP. Σχεδόν το έχουμε πετύχει ε, αυτό το διπλό στόχο. Αλλά δεν το έχουμε κατοχυρώσει ακόμη και θέλω να σας περάσω αυτό το μήνυμα, Υπουργή ότι ακόμη δεν υπάρχει. Ας μην ανοίξουμε σαμπάνιες ακόμη. Έχουμε ε, δουλειά ακόμη για να περατωθεί η διαδικασία και να ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Όπως είπε η σκιώδησε της ομάδας μας που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα δυστυχώς, ποιότητα, όχι μόνο ταχύτητα, Ε, σας παρακαλούμε ε, χρησιμοποιήστε τις τελευταίες ώρες της Ισπανικής Προεδρίας ούτως ώστε ε, να κλείσετε τη συμφωνία. Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Ευχαριστούμε κυρία Ιντβελντ. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε χρόνο γιατί αναβλήθηκε το θέμα TFTP και PNR και η καταστάση επιβατών. Τέλος πάντων, για το TFTP. Είπατε ότι έχει αλλάξει, τροποποιηθεί άρδινη συμφωνία. Θα διαφωνήσω εγώ. Η ουσία ποια είναι η μεταφορά των χίδιν δεδομένων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Θα τα μεταφέρουμε χίδιν ή θα μεταφέρουμε μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται για την ε, διερεύνηση κάποιων ε, υποθέσεων. είναι απλά τα πράγματα. Οι Αμερικάνοι θέλουν ε, θέλουν τα πάντα. Εμείς τι θα κάνουμε, θα του στείλουμε τα πάντα ή θα του, και θα ψάχνουν μόνο τους μέσα στα χείρα ή εν πάση περιπτώσει θα του στείλουμε μόνο ό,τι χρειάζεται και τίποτα παραπάνω. άλλο βέβαια η μεταφορά των χείρων δεδομένων και άλλο η συλλογή του ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αν λέτε ότι δεν υπήρχε απέτηση μέσα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τρία ή για πέντε χρόνια, ξέρετε γιατί έγινε αυτό, διότι θέλαμε να μεριμνήσουμε ώστε να συλλέγουν τα δεδομένα εδώ, στο, ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, είτε χρειαστούν ε, δύο, τρία, πέντε χρόνια, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πέντε χρόνια. Δεν είμαι πεπισμένη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να δεχτώ τα πέντε χρόνια. Είναι δυσανάλογα μεγάλη περίοδος. Υπάρχει και αρνητική μελέτη του EDPS για αυτό το θέμα Τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη, η Γερμανία και το Βέλγιο, επίση ε, συμφωνούν μαζί μου ότι είναι δυσανάλογα μεγάλη περίοδο ε, των πέντε ετών. Ε, για τι καταστάσει επιβατών, λίγα πράγματα θα πω γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Πρώτον για το χρονοδιάγραμμα και τώρα στρέφομαι προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν κρίνετε ότι δεν μπορείτε να τηρήσετε την προθεσμία για τη 15η Ιουλίου για το πακέτο PNR, ε, ίσως υπάρχει σοβαρό σοβαρός λόγος, εν πάση περιπτώσει, για να αναβληθεί. εν περιπτώσει να έρθει να εξηγήσετε γιατί δεν μπορείτε να την την προθεσμία. Δεύτερον, θέλω να ακούσω και από το Συμβούλιο για την Επιτροπή το εξή. Έγιναν σημαντικότερε αλλαγέ για την εφαρμογή ε, τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, τη αμερικανική νομοθεσία ε, για τα ιδιωτικά δεδομένα που επηρεάζουν και του Ευρωπαίου πολίτε. Τι εσεί τι κάνατε, κάνατε νομική αξιολόγηση της κατάστασης. Ε, μία γνωμοδότηση που έχω δει εγώ ε, συνεπάγεται ότι αλλάζει σε μεγάλο βαθμό η, κατάσταση. Τώρα για τα πρότυπα PNR. Γιατί δεν εκπροσωπήθηκε η Ευρωπαϊκή ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση που έγινε, γιατί δεν μας προσκάλεσαν. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας, τι έγινε σε αυτή τη συνεδρίαση. Ο κύριος Κοέλιο, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την συνεργασία που είχαμε με την Ισπανική Προεδρία. Ήταν ε, πολύ χρήσιμα αυτά ε, που έκαναν οι συνεργάτες σας ε, ήταν ακριβής και μεθοδική στις επαφές μαζί μας και διεξοδικά μας ενημέρωναν πιο διεξοδικά σε σχέση με το παρελθόν για τις βάσεις δεδομένων ΔΕΗ ή για το ΣΥΣΕ 2 ποτέ η Προεδρία δεν παρέλειψε το να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Και έτσι κλείσαμε και το, θέμα των θεωρήσεων μακράς διαρκείας και τη μετανάστευση των δεδομένων του ΣΥΣ. Ε, τώρα, για το θέμα της Ρουμανίας και για της Βουλγαρίας δεν είναι λάθος ε, της Προεδρίας, ε, μάλλον του Συμβουλίου, ε, διότι είναι απερίγραψη σχέσεις και συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Μας προκαλούν και είναι η πρόκληση αυτή η επιστολή που έστειλαν για τη Ρουμανία και την Βουλγαρία. Δεν μας ενημέρωσαν συγκεκριμένα, τέλος πάντων το Υπερβήκαμε αυτό χάρη στον πρέσβη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Πέραν αυτού του μεμονωμένου περιστατικού ήταν πολύ θετικά τα αποτελέσματα της Ισπανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε η κυρία Γιγιόμ. Μάλιστα, Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα του ασύλου. Επιτρέψτε μου για λίγα λεπτά αναγνωρίζω ότι έκανε σοβαρό έργο η Ισπανική Προεδρία, αλλά πέρα από την έγκριση για το κοινό γραφείο υποστήριξη για το άσυλο, ε, ουσιαστικά δεν προχώρησαν οι συζητήσει στο Συμβούλιο καθόλου για το πακέτο ασύλου. Ε, Προσπάθω να είμαι σύντομη και θα τα πω συνοπτικά. Ε, ζητώ συγγνώμη. Ε, γιατί παρεμποδίζεται η πρόοδο, διότι οι μηχανισμοί που προβλέπονται, παραδείγματο χάρη για τι διαδικασίε υποδοχή, οι διατάξει λοιπόν συνεπάγονται υπερβολικά μεγάλο διοικητικό άκθο για να χειριστούμε τα άτομα αυτά, για να τι αιτήσει του, να τι επεξεργαστούμε κτλ Μάλιστα, εντάξει, το δέχομαι αυτό το επιχείρημα, αλλά όχι ότι αιτιολογεί και τον περιορισμό ε, των χορηγήσεων ε, ασύλου. Θελήσατε να κλείσετε κακήν κακός κάποια ε, ζητήματα ε, και εσείς ε, προτάσετε το επιχείρημα ότι είστε ρεαλιστές και ότι δεν, να, δεν μπορείτε να σημειώσετε πρόοδο σε όλα τα επιμέρους σημεία του πακέτου ασύλου. Μα συγγνώμη σας ρωτώ, μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για ένα πακέτο ασύλου. Είναι αλληλένδετες οι νομικές αυτές τις πράξεις. Υπάρχει συνοχή ανάμεσα σε όλα τα επιμέρους σημεία. Και για να μην υπερβώ το χρόνο αγόρευσης, να πω και κάτι τελευταίο. Ε, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία και την ε, υποδοχή, δηλαδή σε αυτό τον αιώνα ή τον επόμενο θα πρόκειται να σημειωθεί κάποια πρόοδος και ε, κατοχυρώνεται με κάποιο τρόπο ο έλεγχο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Ο, η κυρία Κέλλερ. Θα δώσω τα δύο λεπτά στο συνάδελφο, απλώ ε, θορυβούμε. Δη, ε, δηλώνω δυσαρεστημένη διότι δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε το άσυλο. Έχουμε μπερδέψει αυτά τα δύο σημεία της σα διάταξη και τελικά δεν συζητάμε τίποτα. Ε, για το TFTP στα γερμανικά. Ich bin ein bisschen überrascht über die Antwort des Rates jetzt zu. Συγγνώμη, αλλά με ξάφνιασε η απάντηση για το TFTP από πλευρά του Συμβουλίου. Δηλαδή, τι, δεν ακούτε πρώτη φορά για την τριετή προθεσμία. Εξ αρχής στο Κοινοβούλιο ε, είπε ότι η μαζική ε, διαβίβαση δεδομένων χίδιν ε, δεδομένων ε, δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο και θέλουμε να βρούμε μία λύση για να ε, παρεμποδίσουμε την μαζική μεταβίβαση δεδομένων. Θέλουμε να γίνεται η έρευνα με στοχευμένο τρόπο για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είχαμε πει εξ αρχή ότι μόνο με συγκεκριμένη προθεσμία θα ε, προσυπέγραφε τη συμφωνία αυτή το Κοινοβούλιο. Σε όλες τις ε, διεθνείς συμφωνίες έχουμε τα χρονοδιάγραμματα, τους όρους υλοποίησης της συμφωνίας, μα γιατί λέτε ότι είναι ανέφικτο να ορίσουμε την προθεσμία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχουμε μια δεσμευτική προθεσμία για αυτή την ε, μεταβίβαση δεδομένων. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε στοχευμένες ε, διαβιβάσεις ε, και να ε, εγκαταλείψουμε την ιδέα της μεταβίβασης. Ευχαριστούμε ο κύριο Σάλβαρο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ για τις απαντήσεις που δώσατε. Νομίζω ότι ε, από τις αντιδράσεις ε, των συναδέλφων ε, θα καταλάβετε ότι δεν είναι κάτι καινούριο για μας αυτό. Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωραία, καλή ιδέα, αλλά εμπεριέχεται ήδη στη συμφωνία. προβλέπεται στη συμφωνία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει και θα αξιολογήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ένα ισοδύναμο πλαίσιο TFTP για την συλλογή των δεδομένων. Τέλος πάντων αναφέρεται αυτό ήδη στη συμφωνία. Επικάλυψη είναι, αλλά ε, εντάξει, καλό είναι που το επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πέντε χρόνια διαφωνώ. Η ίδια συμφωνία δεν εκπνέει μετά από αυτή την προθεσμία. Στα πέντε έτη αυτομάτως παρατείνεται Αυτομάτως παρατείνεται, συνεχίζεται δηλαδή. Εάν είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο, ότι ε, ένα από τα δύο μέρη θέλουν να καταγγείλουν τη συμφωνία, το, ε, τότε περιτεύει το 21-2. Τι λέει το 21-2, ότι ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα έρθετε εσεί και μας πείτε ότι έχουμε σοβαρούς λόγους για τους οποίους θέλουμε να πάυσει η συμφωνία, καταγγέλουμε τη συμφωνία. Ε, στο 21.2 δεν προβλέπεται καμία παραβίαση, στο 21.1 ναι, αλλά ε, το 21.2 δεν αναφέρει όρους, μόνο αυτή την εξάμεινη προειδοποίηση, τίποτα άλλο. Ε, διαφωνώ λοιπόν για αυτό το θέμα και τονίζω και πάλι την απροθυμία που υπάρχει αυτά τα τρία χρόνια και μας λένε ε, τα, αν πιστούν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούμε να έχουμε έναν μηχανισμό συλλογής δεδομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια μέσα σε αυτή την προθεσμία ε, των τριών ετών, δεν θα κάναμε καν αυτή τη συζήτηση προτάσσοντας νομικά επιχειρήματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει βούληση για να γίνει αυτό. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω ε, γιατί υπάρχουν τόσε πολλέ ε, δυσκολίε ε, για να ορίσουμε σαφώς την ημερομηνία ή ένα σαφέ χρονοδιάγραμμα, ούτω ώστε στην τωρινή θητεία του το Κοινοβούλιο να μπορέσει να παρακολουθήσει τη διαδικασία, γιατί είναι δική του αρμοδιότητα. Τρία χρόνια λοιπόν. και όταν όλοι συνεργάζονται μαζί μας και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους, αλλά όταν οι άλλοι είναι απρόθυμοι και εμείς θα είμαστε απρόθυμοι. Ευχαριστούμε, κυρία Λάτφορντ. Πρόεδρε, με τα χαρά συμμετείχα στις ε, επιτυχείς διαπραγματεύσεις ε, για την οδηγία με την Ισπανική Προεδρία για την Ερπινία και ο, ο εκπρόσωπος της Προεδρίας κάθε στα αριστερά σας, Υπουργέ. Υπήρχε πολύ μεγάλη πιστοσύνη ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα και στέφθη με επιτυχία η διαδικασία. Όλοι φύγαμε νιώθοντας ότι είχαμε κερδίσει κάτι, ότι είχαμε νικήσει. Αλλά ε, ας κάνουμε τον παραλληλισμό με αυτή τη διαδικασία για το SWIFT. Είναι το αντίθετο. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη. Ε, και θορυβούμε από την κατάσταση. Μάλιστα, ωραία, έχουν σημειωθεί βελτιώσεις ε, από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα αλλά αυτό ε, οφείλεται ε, συνολικά σχεδόν στο κοινοβούλιο. Μα ποιο είναι το πρόβλημα και ε, γιατί δημιουργούν προβλήματα. Εσείς υπερασπίζετε την οδηγία του Συμβουλίου του 95. Μα δεν ίσχυε η συναπόφαση τότε. Ήταν οδηγία του Συμβουλίου και αυτήν υπερασπίζεστε. Μα, και, εσύ, και μας λέτε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Το πρόβλημα όπως και ε, στο παρελθόν δεν είναι με τη ΣΥΠΑ, είναι με τα άλλα θεσμικά όργανα. Τέλος πάντων ε, έχω και τα ερωτηματικά μου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν αντισχολιάσω. Αλλά το Συμβούλιο σαφώς είναι απρόθυμο. Ακούσατε τώρα τον εισηγητή. Μα δεν ξέρω αν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε, αλήθεια. Ε, είναι φοβερό που δεν μας βοηθάτε ούτω ώστε να έχουμε ένα συνεχές, ε, συνεχή ιστό, μια ομοιόμορφη ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τη ΣΥΠΑ για την καταπολέμηση της ε, οργανωμένης εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Καλή συμφωνία, αλλά είναι ατελής. Η Europol, ε, ε, λέμε, ουσιαστικά θα ευθύνεται για όλα. Μα η Europol έχει συμφέρον για αυτά τα δεδομένα και θα, δεν μπορούμε να τη βάλουμε και υπεύθυνη να την επιφορτήσουμε με την παρακολούθηση ε, της ε, χρήσης των δεδομένων. Και ποιος θα είναι αυτός που μας εκπροσωπεί στη ΣΥΠΑ, θα είναι ανεξάρτητος, θα εμπλέκεται το Κοινοβούλιο στην εκλογή του. Μιλήσατε επίσης για τη μελέτη DPS ότι ήταν αρνητική και είπαν ότι όχι, δεν συμφωνούν με τα πέντε έτοιμα. Εκείνοι μίλησαν για σύντομη μεταβατική περίοδο. Ε, και στην Ω συνήθω ε, κάνει σοβαρέ και δικαιολογημένε επικρίσει ο κ. Χάστινγκ, ο Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία των Ηνωμένων. Αλλά, συγγνώμη, το βάρος πέφτει πάνω σας. Εάν είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος ε, Άλβαρο, τον Αμερικανό πρέσβη, χτες το βράδυ, αμέσως θα του είχατε απαντήσει στο τηλέφωνο, είμαι σίγουρη. Ε, ε, θέλουμε να βελτιώσουμε αυτή τη συμφωνία ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Αν συνεχίσετε να έχετε αυτή την συμπεριφορά μαζί μας, δεν θα τα πάμε καλά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας και για την Ισπανική Προεδρία. Ε, όταν παρουσιάσατε το πρόγραμμα εργασίας ε, δεσμευτήκατε να προστατεύσετε τα θύματα της τρομοκρατίας και να ασχοληθείτε μαζί τους. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι δεν κάνατε αρκετά. Μόνο το ε, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας των θυμάτων. Πολύ καλό είναι και αξιέπαινο, αλλά τελικά εκεί εντάσσονται μόνο οι γυναίκες που είναι ε, θύματα βίας ε, του φίλου. Πολύ καλό αυτό, αλλά δεν έχει να κάνει με την τρομοκρατία. Εμείς θα περιμέναμε, η χώρα μας έχει ταλαιπωρηθεί από την τρομοκρατία, να έχουμε ειδική ε, πρόνοια για προστασία των θυμάτων από τη δρομοκρατία. Χρειάζεται σαφή στρατηγική από τους κυβερνώντες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και δύο φορές είπατε κάτι που με ανησυχήσετε. Είπατε με σθένος και με ανοχή αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατία. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό. Ανοχή, τι ανεκτικότητα. Ποια ανεκτικότητα μπορούμε να έχουμε απέναντι σε εκείνους που δολοφονούν παιδιά αδιακρίτως, πυροβολώντας και με εκρηκτικά και με βόμβες. Υπάρχουν όρια και στην ε, ανεκτικότητα και στην ανοχή. 200 χρόνια ε, μετά τη Γαλλική Επανάσταση ε, αυτά παραμένουν ενισχύ. Δεν συμφωνούμε με αυτό που είπατε. Δεν μπορούμε να ενδίδουμε στους τρομοκράτες και να έχουμε πολιτική υποστήριξη. Δεν μπορούμε να έχουμε διεθνή υποστήριξη απέναντι στους τρομοκράτες. Αυτό επιζητούν εδώ και καιρό από τα θεσμικά μας όργανα. Έτσι. Μηδενική ανοχή και πυγμή και σθένος. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε προ αυτή την κατεύθυνση και με τη ΣΥΠΑ και με όλε τι χώρε που είναι στη δική μα κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο Λόπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από δύο ώρε και ένα τέταρτο τη ενδιαφέρουσα συζήτηση. πραγματικά ε, έχει ακόμα ισχύ η ερώτησή μου. Δεν έχω καλυφθεί νομίζω. <coughs> υπηρεσίες πληροφοριών και ε, οι διοκτικές ε, αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργάζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όταν έγινε η απόπειρα, μάλλον αποσοβήθηκε η απόπειρα του Νιγηριανού ε, στο αεροπλάνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 16 υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας της Ηνωμένων Πολιτείας των ΗΠΑ ομολόγησαν την αποτυχία τους και χρειάστηκε ένας πολίτης να ε, παρεύει για να σταματήσει ε, την απόπειρα. Και στην 11η Σεπτεμβρίου είχαν ε, παραδεχτεί οι Αμερικανοί ότι απέτυχαν οι μυστικές τους υπηρεσίες. Βεβαίως κάνουν την αυτοκριτική τους, αυτό δεν το παραγνωρίζει κανείς. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε καλό συντονισμό στις δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρώπη πληροφοριών και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών και έρευνας για να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο συντονισμός μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Και αν δεν υπήρχε, δεν θα είχαμε ένα σύστημα προειδοποίησης έγκαιρης για να προλαμβάνουμε ε, απόπειρε που ακόμα μπορεί να διεξάγονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τέτοιου είδους εργαλεία όπως το TFTP στην Ευρώπη ή η λίστα ε, με τα δεδομένα των επιβατών που είναι παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και των βασικών εγγύσεων και ελευθεριών θα πρέπει ταυτόχρονα να εξετάσουμε και ένα τέτοιο μέσο, ένα εργαλείο συνεργασίας για τους Ευρωπαίους. Εγώ καθόλου δεν αφισβητώ τα όσα είπε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Αλλά αυτό που είναι γεγονός είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν επίγνωση ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών ε, χρειάζονται μεγαλύτερο συντονισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν την αίσθηση οι πολίτε ότι δεν συντονιζόμαστε αρκετά. Mm. Στο ΚΟΣΙ, λοιπόν, στην Επιτροπή Εσωτερική Ασφαλεία, υπάρχει δυνατότητα τα στοιχεία αυτά τα οποία συλλέγονται ε, τη χάνουν κάποια κεντρική επεξεργασία, κάποιου συντονισμού ή όχι. Η Ισπανική Προεδρία αυτού του μήνε έχει να παρουσιάσει συντονισμό και βελτιωμένη συνεργασία για να μπορέσουμε ακριβώς να αξιοποιούμε τέτοια συστήματα αναλογικά στην καταπολέμηση. Ο κύριος Λαμπρινίδης, τελευταίος. Ξέρουμε ότι μπορεί να είναι σύντομος. No, look. quickly on... Uh, Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για το SWIFT. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες υποστηρίζουν το αίτημα για τα τρία χρόνια το Συμβούλιο ας κάνει ό,τι μπορεί αυτές τις τελευταίες ώρες ε, των διαπραγματεύσεων για να καταλήξει σε συμβιβασμό. Συμφωνούμε με τον κύριο Μπούσελτη. Είμαστε πολύ κοντά. Μπορεί να κλείσει η συμφωνία, αν υπάρξει καλή βούληση από πλευράς όλων. Και έχουμε κάνει ήδη πολύ δρόμο και ευχαριστώ την Ισπανική Προεδρία. Ε, όλοι αγωνιζόμαστε, αλλά δεν πρέπει να, ε, να αναγνωρίζουμε όταν χάνουμε, αλλά ας μην τρεπόμαστε και όταν κερδίζουμε. Και συγγνώμη, το Κοινοβούλιο έχει νικήσει. Όχι μόνο από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά ε, και από τους Αμερικάνους. Στο παρελθόν καν είχαν φανταστεί ότι θα δεσμεύονταν κατά αυτόν τον τρόπο μέσα σε μια συμφωνία. Τέλεια δεν είναι αυτή η συμφωνία σε καμία περίπτωση και ανησυχώ όπως και οι συνάδελφοι για αυτό το θέμα της Europol. Δεν νομίζω ότι τώρα γίνεται να αλλάξει αυτό και δεν θα το ζητήσω ως εκ τούτου. Αλλά θέλω να αναγνωριστεί σαφώς, όπως ε, το λέει στη γνωμοδότησή του και ο κύριος Χάστινγκς, ότι είναι ενιολογικό το θέμα, αλλά και νομικό. ρωτώ το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Τζόναθαν Φόλης και τους άλλους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αν υπάρχει ένας τρόπος και μπορούμε να το συζητήσουμε ώστε όσο η Europol παραμένει το αρμόδιο για την παρακολούθηση όργανο θα εποπτεύεται ε, κατά το δέον. Τι εννοώ. Εάν καταφέρουμε να βάλουμε εμείς σε κάποιον Ευρωπαίο εντεταλμένο στο Υπουργείο Οικονομικών ε, τον ΗΠΑ για να παρακολουθεί τις έρευνες, έτσι μπορούμε να ζητήσουμε κάποιος από, ε, που θα εκπροσωπεί τον Ευρωπαίο Επόπτη προσωπικών δεδομένων να παρακολουθεί την Europol ενώ επιτελεί το έργο της. Αν το καταφέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάλι τέλεια δεν θα είναι η συμφωνία, αλλά θα διασκεδάσει πολλές από τις ανησυχίες που υπάρχουν. Ευχαριστούμε. άλλε ε, δύο παρεμβάσει. Ε, ο, ο κύριος Πίτερ Χάστινγκς, Ευρωπαίος ε, Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μετά ο κύριος Φόλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Χάστινγκ, δύο λεπτά σα παρακαλούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, πολλά μέλη της Επιτροπής ε, παρέπεμψαν στην γνωμοδότηση που υπέβαλα πριν από λίγες μέρες. Εκεί τονίζω ότι έχουν ε, σημειωθεί σημαντικότατες βελτιώσεις, αλλά ταυτόχρονα υπολείπονται σημαντικότερε και ανησυχίες που σχετίζονται με θέματα που δεν έχουν ρυθμιστεί και ανησυχίες που σχετίζονται με άλλα νέα ζητήματα. Και για να είμαι ειλικρινής, έχουμε ακολουθούμε μία λάθος κατεύθυνση. Το βασικό ζήτημα είναι τι θα κάνουμε με αυτές τις ανησυχίες και ποια βήματα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Σχετικά με τις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί, υπάρχουν διεξοδικότερες ρήτρες για τα δικαιώματα ε, όσων υπόκειται σε έρευνες. Ωραία, το καλωσορίζουμε, αλλά πρέπει να ε, μπορεί κάποιο να διεκδικήσει τα δικαιώματά του όταν είναι πολίτη τη Ένωση και διαμένει στη ΣΥΠΑ και πρέπει να ακολουθηθούν οι δέουσε διαδικασίε. Υπάρχει σαφή σχέση με τι προϊούσε διαπραγματεύσει ε, σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ΕΕ. Εάν γίνει αν υπάρχει σταθερή σχέση με αυτή την συμφωνία, τότε γίνεται ενδιαφέρουσα αυτή η εναλλακτική λύση. Δηλαδή έτσι θα καλύψουμε μια ατέλεια που προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ε, τώρα, σε σχέση με τις ε, υπολοιπόμενες ε, ανησυχίες, το βασικό ζήτημα είναι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα. Ε, αν υπερβούμε την αρχή τελικά, το, θέμα είναι, το βασικό θέμα είναι η μαζική μεταβίβαση δεδομένων. Ε, σαφής η διάταξη μέσα στην συμφωνία ότι δηλαδή πρέπει να, είναι, να επιμένουμε στη στοχευμένη αναζήτηση δεδομένων αλλά τι στοχευμένο, θα είναι μαζικά τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται όπως έχει τώρα η συμφωνία. Η σύντομη μεταβατική περίοδος θα βοηθούσε, ούτω ώστε να στοχεύσουμε καλύτερα τη διαβίβαση. Ναι, αλλά αν γίνει όπως πρέπει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κοινό μηχανισμό αναθεώρησης. Να άλλη μια αναλλακτική λύση. Ε, πρώτη φορά μετά από έξι μήνες θα αναθεωρήσουμε τη συμφωνία και μετά σε τακτική βάση θα αναθεωρείται. Βάσει αυτού του ε, μηχανισμού ε, θα έχουμε και καλύτερη στόχευση γιατί θα είναι πιο βραχυπρόθεσμη η εφαρμογή. Τώρα, η Europol δεν είναι δημόσια δικαστική αρχή. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και χρειάζεται δικαστική ε, εποπτεία, αναθεω, ε, παρακολούθηση. Ε, και καλωσορίζω τα σχόλια του κυρίου Λαμπρινίδη. τώρα, πέραν του Ατλαντικού, καλό θα ήταν να βελτιωθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης επίση. Μάλιστα, ευχαριστούμε ο κύριο Τζόναθαν Φόιλ τώρα θα μπορούσατε να απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Ίντεβελτ, γιατί απίφθηνε μια ερώτηση στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να πω και κάποια ε, πράγματα για το TFTP για να δώσω απαντήσεις και έχω και ένα πολιτικό μήνυμα από τη Σεσίλια Μάλμστρομ. Ε, λυπάται που δεν μπορεί να έρθει σήμερα το πρωί και θέλει να σας διαβιβάσω εγώ το μήνυμά τη. Ε, φαίνεται ότι ακούσατε τις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ειλικρινά δεν απηχούν την πραγματικότητα. Νυχθημερών δουλεύουμε. Τα τηλέφωνα τα αφήνουμε αναμένα τουλάχιστον μέχρι τα μεσάνυχτα κάθε μέρα τις τελευταίες ημέρες ούτως ώστε να ε, καλύψουμε τα συγκεκριμένα αιτήματα και τις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου. Το ίδιο κάνει η Επιτροπή και η Ισπανική Προεδρία. Ήταν ταπεινωτικό να ξανανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις με έναν ε, αλλοδαπό εταίρο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι. Κανονικά δεν έπρεπε να χρειαστεί ε, να ξανανοίξουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η τροποποίηση του άρθρου 12. Αυτό έχει κατοχυρωθεί. Επειδή εσείς το ζητήσατε συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες σχετικά με το διορισμό του εντεταλμένου της Επιτροπής, μα θα τα ρυθμίσουμε αυτά. Εμείς θα το συζητήσουμε μεταξύ μας όταν φτάσει εκείνη η ώρα. Το ζήτημα κλειδί, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι κατά τη γνώμη μου, είναι η μαζική μεταβίβαση δεδομένων και πώς θα αποφύγουμε το να χρειαστεί μαζική μεταβίβαση. Δεν θέλουμε να τα στέλνουμε αυτά τα δεδομένα, ε, ε, δεν θέλουμε να στείλουμε όλο το άχυρο για να βρούνε τη βελόνα. Αλλά μέχρι να βρούμε αντίστοιχο σύστημα συλλογής των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, άλλος τρόπος δεν υπάρχει για να ε, λειτουργήσει σύστημα παρακολούθησης χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Οπότε το ουσιαστικό ζήτημα είναι πότε μπορούμε εμείς ε, να ε, συγκροτήσουμε ένα ισοδύναμο σύστημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εσείς το ξέρετε. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα το αποφασίσουν αυτό. Χρειάζεται χρόνος χρήμα ε, και ε, ε, πολλά εκατοντάδες τεχνικά γεωπολιτικά ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν. Εμείς έχουμε αναλάβει μέσα σε ένα χρόνο να υποβάλουμε μια πρόταση, δηλαδή γρήγορα και θα την υποβάλουμε. Η συμφωνία διαρκεί πέντε χρόνια και στις τελικές της διατάξεις αναφέρει ότι ε, οδηγεί, μετά την εκπνοή των 5 ετών ε, ανανεώνεται αυτόματα η συμφωνία εκτός αν υπάρξει καταγγελία από ένα συμβαλόμενο μέρος ε, και συνεχίζεται λοιπόν η συμφωνία βάσει των όρων που η ίδια προβλέπει. Ωραία. Δεν μπορούμε να εισέλθουμε μέσα σε μια, ε, να προσυπογράψουμε μάλλον μια πενταετή συμφωνία και να πούμε στον, στο άλλο συμβαλόμενο μέρος και στον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν θέλουμε τελικά πενταετή συμφωνία, θέλουμε συντομότερη. Μα ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Το Συμβούλιο και αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα της Σεσίλια Μάλθρομ, εγώ είμαι υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο, δεν θα σας εγώ διαβιβάζω μόνο το μήνυμα της κυρίας Μάλστρομ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εδώ πέρα διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία και το Συμβούλιο θα την υποβάλει για την ε, σύμφωνη γνώμη σας. Εσείς ε, βέβαια έχετε την αρμοδιότητα να, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή όχι. Είναι η αρμοδιότητα που σας αναγνωρίζετε μέσα στη συνθήκη. Ελπίζουμε ότι στις 7 Ιουλίου θα υπερψηφίσετε την πρόταση. Τίποτα δεν θα αλλάξει ε, το Σεπτέμβρη σε σχέση με σήμερα. Ε, λοιπόν, μπορώ να μιλήσω μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να σας πω και το κλίμα που επικρατούσε στην Κορεπέρ χτες, γιατί ήμουν εκεί. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε ε, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Ε, ωραία, τώρα υπάρχει αυτό το ζήτημα της διάρκειας της συμφωνίας. Μα αυτό προβλέπεται μέσα στη συμφωνία και είναι άλλο θέμα. Ε, είναι ξεχωριστό σε σχέση με τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού TFTP. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση μέσα σε 12 μήνε να ε, κάνει νέα πρόταση και θα το κάνει. Από εκεί και πέρα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, οι συνομοθέτες δηλαδή θα αποφασίσουν ότι θέλουν να κάνουν. Δεν θα είναι εύκολο να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοθέτημα, αλλά μόλις το κάνετε θα, υπάρχει, θα υπάρχουν διάφορες συνέπειες. Αλλά ας μην ε, το κάνουμε ολόκληρο θέμα. Ε, είχαμε εντολή, διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και, τα, και οι δύο πλευρές της διαπραγματεύσεις και η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική καλόπιστα κινήθηκαν. Ας μην αμφιβάλλετε για την καλή πρόθεση της Επιτροπής. Σταύρο θα σου απαντήσω και μετά θα ασχοληθώ με την ερώτηση της Σόφη Ιντβελ. Παρακαλώ βιαζόμαστε πάρα πολύ. Ωραία. Ε, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Ε, τότε να απαντήσω γραπτό ε, για το PNR, γιατί θέλω πέντε λεπτά για να απαντήσω. Είναι σοβαρό το θέμα. Ε, Είναι πολύ απλό. Μπορώ να απαντήσω λοιπόν μόνο στο Σταύρο. Η Europol. Ε, κοινό εποπτικό όργανο υπάρχει στη Europol για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. Δεύτερον, ε, ως απόρρια αυτής της Διεθνούς Νομικής Συμφωνίας, το δικαστήριο θα έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται για τις δραστηριότητες της Europol στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Οπότε μην ισχυρίζεστε ότι δεν ελέγχει κανείς τη Europol. Έχει την διαχειριστική δομή, έχει το κοινό εποπτικό όργανο ε, όπου υπάρχουν ε, αξιωματούχοι που ελέγχουν ε, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και υπάρχει και απότατη αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της ευρωπαϊκή Ένωσης. Οπότε μη μου μιλάτε για τη λισαβονοποίηση του ρόλου της Europol. Αυτά συνεπάγει για τη λισαβονοποίηση. Ε, Σοφή, συγγνώμη, έχω πλήρη απάντηση να σου δώσω, αλλά θέλω πέντε λεπτά. Πρόεδρος, Επιμένει η κυρία Ιντβέλτ ε, να πάρει απάντηση γιατί θα πάει με το κλιμάκιο στη ΣΥΠΑ για τα θέματα ε, των καταστάσεων επιβατών και θέλει την ε, απάντηση. Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα. Και από πλευρά των συναδέλφων σχεδόν εισηγητών. Ωραία, θα δεχτούμε τη γραπτή απάντηση, αλλά τη θέλουμε μέχρι αύριο, γιατί φεύγουμε για την Ουάσιγκτον για τα θέματα PNR. Μέχρι το γεύμα θα την πάρετε. Ακόμη καλύτερα. Τονίζω ότι επανειλημμένα έχουμε υποβάλει γραπτό σε αυτά τα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποτέ δεν πήραμε απάντηση και γι' αυτό και το συζητάμε σήμερα. Το εγγυώμαι, θα σας έρθει η απάντηση. Ωραία, να πω και με ένα προσωπικό σχόλιο, κλείνοντας την παρέμβασή μου. Τελευταία φορά έρχομαι στην Επιτροπή σας όντως, Πρόεδρε. Με την τωρινή ιδιότητά μου, πραγματικά η εφροσύνη των μελών της Επιτροπής σας ε, ενώπιον μου ήταν ανέκαθεν καταπληκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Φόλε, εκτιμούμε πολύ ε, τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Πολύ βρετανική συμπεριφορά από πλευράς του κύριου Φόιλ ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής το αφιέρωσε σε αυτό το φάκελο και λυπούμεθα και εμείς πολύ που θα αποχωρήσει, λέει ο κύριος Λαμπρινίδης. Μάλιστα, ε, εκτιμούμε τα όλα όσα κάνατε Ευχαριστούμε κύριε Τζόναθαν Φόιλ, σας ευχαριστώ εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Η κυρία Ίντεβελ θα πάρει την απάντηση πριν το μεσημεριανό γεύμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να φάει, αλλά μέχρι το γεύμα, την ώρα του γεύματος, θα έχει πάρει την απάντηση. Ε, ε λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο σημείο. Τώρα θα τα απαντήσει όλα μαζί ο κύριο Ζουμπακάλμπα, ο Υπουργό. Κοιτάξτε δείτε, είμαστε πίσω σε σχέση με το χρονοδιαγραμμά μας. Όμως, συζητήσαμε και όχι για πρώτη φορά αυτό το τόσο επιμαχό θέμα, το τόσο σημαντικό, τόσο λεπτό. Οπότε παρακαλώ θα πρέπει να δείξετε κατανόηση και ε, τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε την καθυστέρηση αυτή. Γιατί ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ο Προεδρεύων του Υπουργείου Δικαιοσύνη περιμένει, περιμένει να έρθει η ώρα του να μιλήσει και αυτό μαζί μα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο γιατί ο κύριος ε, Φολ με, με εκάλυψε ως επιτοπλίστων σε αυτά που ήθελα να σας πω για την Europol, για τον δικαστικό έλεγχο, γιατί ακριβώς μια διεθνής συνθήκη τροποποιεί εν μέρει τον ε, κανονισμό της Europol, οπότε ακριβώς ε, λειτουργώντας η Europol υπό την αιγίδα αυτήν την διεθνή, ε, υπόκειται και αυτή στην τροποποίηση του κανονισμού της Οργανισμού λειτουργία τη πρώτον. Φυσικά και σημειώσαμε βήματα προόδου, ουδή, εξ όσων έλαβαν το λόγο παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι η συνθήκη που έχουμε στα χέρια μας ε, διαφέρει από εκείνη την οποία απέρριψε το Κοινοβούλιο πριν από κάποιους μήνες. Επομένως, ναι, υπήρξαν βήματα πρόοδου. Αρκετά δεν ήσαν αρκετά. Αυτό είναι υποκειμενικό. Πάντως όλα τα θεσμικά όργανα προσπαθούμε να ακούσουμε τη γνώμη των άλλων ε, το ίδιο ισχύει και για η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι χθε το βράδυ είχαμε εξελίξεις γιατί είχαμε τις τελευταίες πινελιές σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου χθε βράδυ στην Κορεπέρ μέσω αυτών των επαφών Συμβουλίου και Κοινοβουλίου τον κύριο Άλβαρο που είναι ο εισηγητής σας επομένως ισχύει το ότι δεν καλύψαμε 100% όπως είχαν ζητηθεί, αλλά αυτό το οποίο ισχύει ότι η χθεσινοβραδινή απόφαση του Συμβουλίου καλύπτει αυτό το άρθρο ή στο οποίο θεσπίζεται υποχρέωση νομικά δεσμευτική τη Επιτροπή, ούτω ώστε μέσα σε ένα χρόνο να παρουσιάσει τι προτάσει τη, ούτω ώστε να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για να ρυθμιστεί το θέμα του SWIFT ή στην Ευρώπη. Αυτά στο άρθρο 2. Στο, στο άρθρο 3 λέει για μία ε, πενταετία κατά την οποία θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία συμφωνία ή να παρούμε σε αναθεώρηση τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Οπότε θα πρέπει σε αυτή την περίοδο να αποφασίσουμε για το κατά πόσο θα προχωρήσουμε ή όχι. Και άμα δεν προχωρήσουμε, τότε θα πρέπει να ληφθούν οι δέουσε αποφάσει. Άρα είχαμε αλλαγέ μέχρι και χθε το βράδυ. Δεύτερον. Όχι. Δεν είμαστε κατά ως Συμβούλιο του να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό SWIFT. Όσον αφορά αυτή τη μαζική διαβίβαση δηλαδή που έχετε τις αντιρρήσεις, η εναλλακτική, η λύση είναι αυτή. Να υπάρχει επομένως μια τέτοια μεταβατική μορφή, ούτω ώστε να υπάρχει ο έλεγχος σε σχέση με το να μην υπάρχει εκτροπή σε αυτή τη ε, διαβίβαση των δεδομένων προς τις ίπα. Ε, Όμως αυτό είναι λύση προσωρινή. Η οριστική λύση θα είναι το να μπορέσει η Ευρώπη να έχει το πάνω χέρι σε όλα όπως είπε η κυρία Ινετφέλτ με το παράδειγμα το οποίο μας έδωσε επομένως αυτό είναι δυνατόν να υπάρξει μόνο αν έχουμε ένα ευρωπαϊκό SWIFT, για το οποίο εμείς δεν έχουμε καμία, καμία αντίρρηση. Είμαστε υπέρ του να υπάρξει. Ούτε καν θέλουμε να υπάρξει διοργανική, διαθεσμική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμών οργάνων και έτσι να ε, όσον αφορά μια κατακλητική ημερομηνία μέχρι την οποία να έχει φτιαχτεί το ευρωπαϊκό SWIFT. Έχουμε αυτή την τριετία που έχει οριστεί, οπότε θα το ορίσουμε και μπορούμε να το κάνουμε και φυσικά το Συμβούλιο θα είναι ο τελευταίο που θα πει όχι σε κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε είναι ότι σε αυτή τη συμφωνία να, να υπάρχει ως προϋπόθεση να υπάρχει ως προϋπόθεση η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή να πούμε ότι ναι, θα φτιάξουμε ευρωπαϊκό SWIFT και αν δεν τα καταφέρουμε τότε θα κάνουμε το SWIFT με εσά. Αυτό δεν μου φαίνεται λογικό γιατί τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ είναι με αυτόν τον πενταετή ορίζοντα δεν είναι δυνατόν επομένω να βάλουμε ως προϋπόθεση τη διοργανική συμφωνία. Επομένως, ναι, να υπάρξει το ευρωπαϊκό SWIFT το νωρίτερο δυνατόν. Και γι' αυτό και Ευχαριστώ είπαμε ναι στην πρόταση Άλβαρες και να δοθεί αυτή η εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε να μας παρουσιάσει το πλαίσιο αυτό. Αν θέλουμε να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία σύμφωνη. Να μην τίθεται όμως ως προϋπόθεση του SWIFT, το να τα βρούμε εμείς μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να πούμε στη ΣΥΠΑ ότι εάν δεν τα βρούμε μεταξύ μας. Η ορίζοντας ο πενταετής θα γίνει τριετής. Que sea no a la Αλλιώς, αν θέλαμε να τεθεί με τέτοια προϋπόθεση, θα έπρεπε αυτό να το έχουμε πει με τη ΣΥΠΑ και να πούμε όχι πενταετία αλλά τριετία. Θεμητό είναι το θέλει αυτό κάποιο. Ε, Όμω δεν είναι δυνατόν αυτό να το εξαρτήσουμε από το Ευρωπαϊκό SWIFT. Άρα Συμφωνούμε με την πρόταση του Κοινοβουλίου. Συμφωνούμε με την πρόταση Λάντφορντ. Δεν είναι δυνατόν η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ όμω να εξαρτάται από το αν εμείς θα μπορέσουμε να τα βρούμε. Το να υπάρχει με τέτοια λύση και δέσμευση για την τριετία, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Ας το κάνουμε αυτό επίσημα. Αυτό όμως είναι δικό μας. Δικό μας θέμα δεν έχει καμία σχέση με τη συνεννόηση και δέσμευση προς τη ΣΥΠΑ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος. Σας αποχαιρετούμε. Ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε. Δεν θα διακόψουμε. Έρχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να πει τα σχετικά συμπεράσματα.

Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. We beg you to take your seats. Καθίστε σας παρακαλώ. Como anunciamos y sin dilación. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, σας παρακαλώ καλωσορίζουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνη ε, της Ισπανική κυβέρνηση, κύριο Φρανσίσκο Καμάνιο, που εκπροσωπεί τη εκπεριτροπής ε, Προεδρία του Συμβουλίου σε θέματα δικαιοσύνη. για να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα ε, του εξαμήνου τη Προεδρίας και μετά από τη σύντομη τοποθέτησή του, παρουσίασή του θα έχουμε ανταλλαγή απόψε. Παρακαλώ 15 λεπτά κύριε Υπουργέ, όχι παραπάνω, διότι ο προηγούμενος Υπουργός μας κράτησε πολύ περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει στην αρχή. Για να ακούσουμε μετά τους συντονιστές και ε, τα μέλη, όλα τα μέλη που θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Φρανσίσκο Καμάνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση επανέρχομαι στην Επιτροπή σας για να σας ε, παρουσιάσω τη τον απολογισμό της ε, Προεδρίας. Ήρθα το Ιανουάριο για να σας εξηγήσω το πρόγραμμα εργασίας που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε το εξάμεινό μας και να σας ζητήσω την υποστήριξή σας και τη βοήθειά σας. Επιτρέψτε μου τώρα να ε, σας εκφράσω τη μεγαλύτερη δυνατή μου αναγνώριση και ε, μεγάλες ευχαριστίες για την πιστή και γόνιμη συνεργασία που είχαμε και τολμώ να χαρακτηρίσω σημαντικά τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα για το στόχο που έχουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που να βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθεριών και στην υπηρεσία των πολιτών. Η Προεδρία μας χαρακτηρίστηκε από την έναρξη μιας νέας ε, περίοδου ε, βαθέων ε, μεταρρυθμίσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη και ιδιαίτερα για τον χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. βασικός παράγοντας αλλαγής αυτής, που είναι πολύ μεγάλη με ελληνικούς, ήταν η θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας που συνέπεσε με τη το νέο πρόγραμμα, το πενταετές πρόγραμμα 2010-2014, το λεγόμενο πρόγραμμα της Στοχόλμης στον τομέα των εσωτερικών και της δικαιοσύνης. Και σε εμά έπεσε ο κλήρος να ε, δώσουμε ε, την έναρξη του προγράμματος αυτού. Τελήσαμε η μετάβαση να γίνει με τρόπο συντεταγμένο ε, στη συνεργασία στην ποινική δικαιοσύνη είχαμε ως στόχο να ε, κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές έτσι ώστε να φτάσουμε ε, στην ε, επιθυμητή ταχύτητα πορείας του συντομότερο βέβαια. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου η δεύτερη Επιτροπή Μπαρόσο δεν είχε αναλάβει ακόμα καθήκοντα. Είναι δύσκολη η φάση αυτή γιατί πρόκειται για ένα ροντάρισμα ε, μέχρι να μπει στο νερό, το νερό στα βλάκι ε, για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είχαμε θεσμικές διεκδικήσεις ή ακόμα και διεκδικήσεις αρμοδιοτήτων και εξουσιών που καμιά φορά έκαναν παρεμβολές ε, στην ήρεμη και επικοδομητική επεξεργασία των προβλημάτων ουσίας. Όπως θα καταλάβατε, αναφέρομαι στη θέση που ακολούθησε η ε, Αντιπρόεδρος κυρία Ρέντινγκ ε, απέναντι στις δύο πρωτοβουλίες των κρατών μελών τις οποίες είχαμε υποβάλει στη συνεργασία για τα ποινικά θέματα. Ε, ε, χρησιμοποιώντας κυρίως ε, τις εξουσίες που μας δίνουν οι συνθήκες ε, στη συγκεκριμένη ακριβώς ποινική συνεργασία. Υπήρξαν εντάσεις εντάσεις οι οποίες σε κάποιο βαθμό εμπόδισαν τη λειτουργία της συνεργασίας με τη Νέα Συνθήκη που είναι ε, πολύ σημαντική. Όπως, αυτό είναι τα ειχέγγυα, τα δικονομικά στις ποινικέ υποθέσεις και η προστασία των θυμάτων. Πάντως, με διάλογο, με επιμονή, με αιμονή, με επιχειρήματα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας καταφέραμε όλοι να επενικήσουμε τα εμπόδια. Εδώ είχαμε ανεκτήμητη ε, βοήθεια από τη δική σας Επιτροπή και από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Δημόσια εδώ να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε στη συνέχεια να σας αναφέρω τις σημαντικότερες ε, πρόοδους της περίοδου τούτης που συμπίπτει με την εκτέλεση, όπως σας είπα, της αρχικής φάσης του προγράμματος της Σοχόλμης. Στο Συμβούλιο εγκρίναμε κάποια συμπεράσματα σχετικά λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανα μια σύντομη αναφορά στην αντίστοιχη οδηγία τα δικαιώματα ε, διερμηνίας και μετάφρασης ε, στην ποινική δικαιοσύνη. Είναι το πρώτο νομοθέτημα που εγκρίνεται στα πλαίσια της ε, ποινική δικαστικής συνεργασίας μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Σαββόνας. Σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία κανονική, συνήθη. Επίση, σε πρώτη ανάγνωση πρέπει να τονίσω ότι επέτρεψε τη συμφωνία αυτή. Θέλω να θυμίσω ότι είναι αυτό ένα πρώτο μέτρο του φύλου πορείας, του οδικού χάρτη που όλοι εγκρίναμε στη Σουηδική Προεδρία, έτσι ώστε σταδιακά να περάσουμε από αυτή την τεχνική και βαθμία ε, μέθοδο στην ενίσχυση των ε, ποινικών δικονομικών εγγυήσεων για να ε, αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αρχής της αμοιβαία αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων. Αυτό είναι ακρογωνιαίος λήθος για οποιαδήποτε ε, δικαστική συνεργασία. Αυτή λοιπόν η επιτυχία θα πρέπει να είναι κίνητρο για μας έτσι ώστε αποφασιστικά να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα βήματα του φύλου πορείας ή του οδικού χάρτη αρχής γενομένης από το δικαίωμα ενημέρωσης στο κρατούμενο και προσεχώς περιμένουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι μπορούμε ειλικρινά να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για ε, το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Εδώ είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά η Επιτροπή σας και η συγγήτριά σας Βαρόνι Λάτφορτ όταν αποφάσισε να εργαστεί βάσει της πρωτοβουλίας που από κοινού 13 ε, κράτη-μέλη καταθέσαμε μετά από πρώτερη πολιτική συμφωνία και να μην λάβει ως κείμενο φετηρία στην πρόταση ε, που ευνηδιαστικά έφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιδών Δικαιωμάτων είναι Κάτι το οποίο εναπόκειται στα κράτη-μέλη και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εσωτερικό της Ένωσης σε όλα τα θεσμικά όργανα. Χωρίς κανένα να σφετερίζεται το μονοπόλιο της ερμηνείας. Όλοι ε, θεσμικά μπορούμε να ερμηνεύουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών. Και κανείς δεν επιτρέπεται ε, στη διαδικασία πώλησης ενός προτύπου, ενός κανόνα να αυτό ανακηρύσσεται σε αποκλειστικό θεματοφύλακα. Θα πρέπει όλοι να προχωρούμε προς την ίδια κατεύθυνση με συνεννόηση και ευτυχώς τελικά αυτό έγινε και με την παρούσα οδηγία. Οι συζητήσεις, θυμίζω στην τομία, ε, στράφηκαν γύρω από τρεις μεγάλους άξονες. Την διερμηνία ε, στις ε, συναντήσεις του υπόπτου ή του κατηγορουμένου με το δικηγόρο του, ε, η δυνατότητα μετάφρασης ή ακόμα και η δυνατότητα απόρριψης, άρνησης μετάφρασης. Αυτά τα τρία είναι και θέματα συναπόφασης Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλοι ποντάρουμε ε, σε υψηλό επίπεδο οικονομικών εγγύσεων για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο για να λυθούν και τα διάφορα τεχνικά ζητήματα που ανέκυψαν. Κυρίε και κύριοι, μια από βασικέ βασικές ε, προτεραιότητες της Προεδρία Προεδρίας ήταν, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Σας είχα πει τον Ιανουάριο ότι είχαμε ε, την πρόθεση να φέρουμε το κέντρο βάρους στην προστασία στα θύματα. Όχι μόνο εγγυήσεις για τους ε, ε, κατηγορουμένους ή τους εγκληματίες, αλλά και προστασία για τα θύματα. Καλύτερη προστασία, καλύτερη βοήθεια, καλύτερη υποστήριξη και υπόθαψη, των θυμάτων. Σεμινάριο επίσης ε, σχετικό διοργανώσαμε και ασχολήθηκε και το άτυπο συμβούλιο του Τολέδο. Σκεφτόμαστε πάντα τα θύματα και πώς μπορούμε καλύτερα να τα προστατεύσουμε βάσει των ε, αρμοδιοτήτων που ε, δίνει στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία η συνθήκη κάναμε μια πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκού Εντάλματος Προστασίας μαζί με 11 άλλα κράτη-μέλη. Από την αρχή εργαστήκαμε με επικοδομητικό πνεύμα, συνενετικό πνεύμα, επιζητώντας συμβιβασμού, συνεννόηση και πάντα συνενετικά επαναλαμβάνω. Ήταν περίπλοκο αυτό το εγχείρημα, αλλά και συναρπαστικό. Συγκρούστηκαν δύο απόψεις που κινούσαν από διαφορετικές θεσμικές θέσεις. Η νομική συζήτηση επικεντρώθηκε στην ερμηνεία της έννοιας του ποινικού δικαίου και πώς αυτό προβάλλεται στη συνεργασία των ποινικών δικαστηρίων υπό το φως της συνθήκης Λισαβόνα. Τα περισσότερα κράτη-μέλη, αλλά και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, θεωρούν ότι το σημαντικό για να δούμε το πεδίο δράσης του ποινικού δικαίου είναι το υποκειμενικό στοιχείο που επιτρέπει ε, να δημιουργηθεί αυτόνομο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και όχι τα δικονομικά διάφορα στοιχεία που συνάπτονται στην κάθε διαδικασία και στην κάθε δικονομία που ισχύει στην πραγματικότητα σε κάθε κράτος μέλος. Εμείς Είμαστε υπέρ του αυτόνομου στοιχείου χωρίς το ένα κράτος να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Και η προστασία των θυμάτων να ορίζεται από δικαιοδυτικά όργανα του κράτους μέλους στο ίδιο το κράτος. θα πρέπει στην ποινική νομοθεσία των κρατών ε, και των δύο κρατών ε, να ε, ορίζονται αυτά και να υπάρχει σαφής εικόνα αν έχουμε απειλή ή κίνδυνο για την ελευθερία για τον κατηγορούμενο, για το θύμα. Αλλά τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ περιοριστικά ερμηνεύει τη συνθήκη με χαρακτήρα αποκλειστικά δικονομικών ήθελε να περιορίσει το νομοθέτημα αυτό στην τυπική ε, ποινική διαδικασία εξαιρώντας και αποκλείοντας κάποια άλλα που δεν είναι νόμεν γιούρις ποινικά αλλά έχουν αντίστοιχη φύση ε, λόγω του περιεχομένου, του αντικειμένου, των εγγυήσεων κτλ. Όπως συμβαίνει με κάποιες διαδικασίες όπου οι ε, δικαστικές αρχές ε, υιοθετούν μέτρα προστασίας και εγγύησης των ελευθεριών, για παράδειγμα, στο οικογενειακό δίκαιο. Como estamos también en una política, es... Ε, τώρα όμως, επειδή είμαστε και πολιτικοί, δεν θα πρέπει να αφήνουμε τα φαινόμενα να μας απατούν και θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Δηλαδή, αν σταθούμε λίγο και κοιτάξουμε αυτή την κατάσταση, πίσω από αυτή τη νομική συζήτηση κρύβεται ε, μια διελκυστίδα για το ποιος θα έχει την πρωτοβουλία ή για να το πω με άλλα λόγια. Ένα κίνημα για να περιοριστεί ε, το θέμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το πλαίσιο που είναι καινούριο, είναι νέο έδαφος ε, που εξερευνούμε τώρα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μόνο από αυτήν άλλωστε την προοπτική και το πρίσμα μπορεί κανείς να καταλάβει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προσκολήθηκε, επέμεινε, τα στήλωσε για να ε, διατηρήσει το μονοπόλιο της ε, πρωτοβουλίας ε. μένοντας πάρα πολύ στους τύπους χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής συγγνώμη, των νομικών υπηρεσιών και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προσωπικά μου τράβηξε την προσοχή το γεγονός αυτό ότι επέμειναν πάρα πολύ τόσο τυπικά στην ερμηνεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα τυπικά και επίσημα υπάρχουν μόνο δύο νομικές νομοδοτήσεις, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Τυπικά και επίσημα δεν υπάρχει τίποτα γραπτό από τις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που τόσο τυπική είναι και μένει σε αυτή τη θέση. Ε, το σημαντικό ποιο είναι σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία όμως. Υπάρχει πλέον ομοφωνία ως προς τους πολιτικούς στόχους και τι σκοπό εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Σε όλα τα κράτη-μέλη, και συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό η ίδια, Αλλά εμεί πιστεύουμε, όπω μα είπαν οι δικέ μα νομικέ υπηρεσίε, αλλά και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, ότι υπάρχει επιπλέον και νομική βάση για να προχωρήσει και να δοκιμήσει αυτή η ε, πρωτοβουλία. Αλλά εκτός από αυτή τη νομική βάση και τους νομικούς λόγους, υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι κατά την άποψή μας που συνηγορούν προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή στο θέμα αυτό να εγκαταλείψουμε την προηγούμενη ε, φορμαλιστική, τυπική και περιοριστική στάση μας. Ακριβώς για, για την προστασία των θυμάτων. Και να πούμε in dubio pro δηλαδή ε, σε περίπτωση αφιβολίας είναι υπέρ του θύματος. ειδικά αυτό αφορά τις γυναίκες που ε, είναι ε, θύματα ε, βίας με βάση το φίλο τους για την προστασία των θυμάτων και αυτό θα πρέπει να είναι ένα κίνητρο το οποίο να μας οθεί γιατί ο λόγος ύπαρξης των θεσμικών οργάνων είναι οι πολίτες. Και οι πολίτες ακριβώς που είναι βάλωτε, που είναι θύματα και κυρίω οι γυναίκες που υφίστανται την ενδοοικογενειακή βία και θα πρέπει να αισθάνονται πραγματικά ότι προστατεύονται. Κυρίες και κύριοι, Αυτές λοιπόν ήταν οι πολιτικές σκέψεις και οι πολιτικοί λόγοι και οι νομικοί λόγοι που μας οδήγησαν τον Ιούνιο στο Συμβούλιο Υπουργών να ε, υποστηρίξουμε κατά πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. 18 κράτη-μέλη το υποστήριξαν ε, και είναι ε, αναφορά για το διάλογο στη συναπόφαση. Θα ήθελα τώρα να αφαιρθώ στην ιδιαίτερη κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου που το Μάρτιο ε, δήλωσε ότι θέλει ε, να ασκήσει το δικαίωμα του opt-in και μετά όταν άλλαξε η κυβέρνηση ε, ζήτησε να απέχει από τη διαδικασία αυτή. Θέλει να καθίσει λίγο να το σκεφτεί. Και ζήτησε περίοδο περισυλλογή. Η Προεδρία του Συμβουλίου άκουσε τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και θεώρησε σκόπιμο να απευθυνθεί στο άρθρο 3 ε, εδάφιο 2 στο πρωτόκολλο 21 για τη θέση της Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Βασιλείου στο χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Εδώ ορίζεται πραγματικά μια περίοδος εύλογη για να είναι αδρανές το opt-in με την ε, υπόθεση ότι Ε, δεν θα παρεμποδιστεί η λήψη απόφασης. Με την επιφύλαξη λοιπόν ε, αυτού του άρθρου και μετά ε, από τη γνωμοδότηση των νομικών μας υπηρεσιών, οι Βρετανοί φίλοι μας έχουν προθεσμία μέχρι το επόμενο Συμβούλιο για να συμμετάσχουν, να θέλουν ή να μην συμμετάσχουν σε αυτό το μέτρο, αν συμπαραταχθούν με την πλειοψηφία ή όχι τον κρατών. Τον Ιούνιο δόθηκε πραγματικά αυτή η ερμηνεία που σας είπα, όχι περιοριστική που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό λοιπόν, και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει διαδικασία συναπόφασης, ε, το κοινοβούλιο σας να ε, συνεισφέρει με τρόπο οριστικό και αποφασιστικό ε, στη βελτίωση του κειμένου και στην οριστική του διαμόρφωση. Γνωρίζω ότι αυτό θέλει να κάνει και η επόμενη Προεδρία, η Βελγική, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ε, άλλωστε γι' αυτό με έχει ενημερώσει η κυρία Ρομέρο, η συγκήτριά σας και η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ Σκιώδης η συγκήτρια και δράτω με τις ευκαιρίες για να τη συγχαρώ για το έργο τους. Είναι πραγματικά ε, προσανατολισμένη προς τους πολίτες και τις γυναίκες όλης της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Τον Ιανουάριο σας είχα πει και άλλες προτεραιότητες που είναι η ενίσχυση των θεμελιδών δικαιωμάτων και το άρθρο 6 εδάφιο 2 της Σύνθηκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν και παρά τις πολλές τεχνικές δυσκολίες που γνωρίσαμε, καταφέραμε να εγκρίνουμε την εντολή για διαπραγμάτευση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ΕΣΔΑ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950. Έτσι, εγκαίρως θα ε, ανταποκριθούμε στο πρόγραμμα της Στοχόλμης που χαρακτήριζε αυτό το θέμα και ε, προτεραιότητα και επίγον. Θα ήθελα δημόσια εδώ να ευχαριστήσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την ανεκτήμητη βοήθειά της για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Όταν κατέθεσε στις 17 Μαρτίου την, ε, τη συστάσεις της, είπαμε ότι είχαμε πολύ καλή βάση εργασίας και το είπαμε τότε, το δηλώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, φιλοδοξούσαμε να εγκρίνουμε την απόφαση αυτή κατά τη διάρκεια ακόμα της Ισπανικής Προεδρίας. Προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησε πάρα πολύ η πολιτική όθηση που πήραμε από το Κοινοβούλιο. Στη Ολομέλεια του Μαΐου εγκρίθηκε αντίστοιχη έκθεση του κυρίου Χαόρεγγι. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν τους εισηγητές είναι πολύ καλή η ε, ε, αφετηρία αυτή για τη διαπραγμάτευση που τελικά θα πρέπει να καταλήξει στη συμφωνία προσχώρηση, δηλαδή να προσυπογράψει η Ένωση την ΕΣΔΑ. Πολύ γοργά έγιναν ε, όλα αυτά, αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου εις βάρος της ποιότητας η ταχύτητα. Και έτσι, μέσω εσωτερικών ρυθμίσεων και παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, θα καταφέρουμε να λύσουμε τα δύο τεχνικά ε, ζητημάτα που ήταν τα πιο περίπλοκα και τα πιο δύσκολα. Δηλαδή, τι γίνεται με το μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών με ε, ένωσης με τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να ξέρει ε, ποια από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί ε, να είναι αντικείμενο προσφυγής στο δικαστήριο του Στρασβούργου ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ των προτέρων. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει μια ε, πιστή συνεργασία πάντα από τους εκπροσώπους των 7 κρατών μελών που θα διαπραγματευθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ορίστηκε ως διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, ε, Επιτροπή ε, θα πρέπει να αναφέρει ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το ενημερώνει σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας και στην αρμόδια Επιτροπή και στην ομάδα εργασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων να αναφέρει επίσης και να ενημερώνει. Η έγκριση της εντολής σίγουρα είναι πολύ καλή είδηση για όλους μας και θα ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο του Ιουνίου επίσης συμφώνησε για ε, κοινή προσέγγιση της οδηγίας που έχει σχέση με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το τράφικινγκ και την προστασία των θυμάτων. Είναι μια πρόταση που φιλοδοξεί να ενισχύσει την πρόληψη αλλά και την καταστολή και την τιμωρία τόσο σημαντικών ε, εγκλημάτων που ε, αφορούν και παραβιάζουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Υπάρχει μια παλιά ε, απόφαση πλαίσιο του 2002. Βάσει του κειμένου αυτού θα μπορέσουμε να αρχίσουμε το διάλογο πάλι σε συναπόφαση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για να εγκρίνουμε τελικά αυτό το τόσο απαραίτητο μέσο το συντομότερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταυτόχρονα κατέθεσε και μια άλλη πρόταση με στόχο να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σεξουαλικής ε, κακοποίησης ε, των αλληλίκων και την παιδική πορνογραφία και στο Συμβούλιο δίνεται συνέχεια ε, με τη Βελγική Προεδρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτού του είδους η εγκληματικότητα είναι πάρα πολύ ιδεχθής, ιδιαίτερος ιδεχθής. Κυρίες και κύριοι, ακόμα και αν δεν είναι άμεση αρμοδιότητα της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, επιτρέψτε μου να αναφερθώ, γιατί έχει σημασία για τους πολίτες, στην έγκριση της ενισχυμένης συνεργασίας για πρώτη φορά μεταξύ 14 κρατών μελών για το νόμο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διαζυγίου και χωρισμού δικαστικού. Πολύ σημαντικό βήμα έχουμε κάνει για να δώσουμε απάντηση σε ένα θέμα που απαιτούσε ευρωπαϊκή λύση και ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πάρα πολλούς διασυνοριακούς γάμους πλέον ε, στην Ένωση και ε, θα έπρεπε να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είμαστε σε θέση πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις ε, χωρισμού και διαζυγίου να ορίσουμε ποιος είναι ο κανόνας που πρέπει να ισχύει και πώς θα διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση διαφωνίας. Ε, ε, στο περιθώριο τώρα ε, του νομοθετικού πεδίου, το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης εγκρίναμε απόφαση για μοντέλο συμφωνίας για δημιουργία κοινών ομάδων δίωξης που θα αντικαταστήσουν τις προηγούμενες και θα υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές. Ήταν μια ιδέα της Προεδρίας που την ε, προώθησε μαζί με τη Eurojust με στόχο ακριβώς να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα και να είναι καλύτερα οπλισμένοι ε, στο αγώνα τους κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Το ε, Ιανουάριο σας ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση της Προεδρίας να κάνει μια πρώτη διερευνητική ε, προσέγγιση ε, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα που προβλέπεται στο άρθρο 86 της Συνδίκης της Ένωσης. Να βολιδοσκοπήσουμε την κατάσταση, το συζητήσαμε αυτό τον Απρίλιο ε, με στόχο να προετοιμάσουμε το δρόμο, να προλιάνουμε το έδαφος για μια περισυλλογή τους επόμενους μήνες και έτη. Το πρόγραμμα δράσης του προγράμματος Στοχόνης προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ανακοίνωση σχετικά το έτος 2013. Ως Προεδρία δεν εναπόκειται σε μένα τώρα να προεξοφλήσω θέσεις, αλλά θα ήθελα να ε, πω ότι είναι αρκετά προβληματικό το πλαίσιο για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και ε, το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως το αναφέρει η συνθήκη είναι κάτι που ε, προσλαμβάνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ε, θα πρέπει να διερευνήσουμε τις δυνατότητες Eurojust ως σύστημα που θα πρέπει να προωθήσουμε στην Ένωση. Αξίζει επίση να τονίσουμε τα συμπεράσματα του Ιουνίου για τη βελτίωση της πρακτική εφαρμογής του Ευρωπαϊκού ε, Εντάλματος σύλληψη και παράδοση που εγκρίθηκε πέρσι. Ε, Αξιολόγησαμε ε, την εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη. Αυτά τα συμπεράσματα διευκρινίζουν ορισμένα στοιχεία και κυρίως φέρνουν την πρακτική εμπειρία την ε, πραγματική χρήση στην πράξη του εργαλείου αυτού και επιτρέπουν ε, αξιολόγηση για να το βελτιώσουμε. Στο Συμβούλιο του Απριλίου εγκρίναμε επίσης ε, αρκετά συμπεράσματα για την πρόληψη οικονομικών κρίσεων ή της οικονομικής κρίσης της τωρινής. Αυτό το θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντικό γιατί και από πλευράς δικαιοσύνης μπορούν να γίνουν πάρα πολλά για να βελτιωθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών για να δούμε και από ευρωπαϊκή σκοπιά για αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν ασχοληθήκαμε με ζητήματα που έχουν να κάνουν. Για το πώς θα φτηνένουν η διαδικασία και η πρόσβαση σε... Το εκτελεστικό της απόφασης. Να καταργηθεί το εκτελεστικό της, της απόφασης για να είναι πιο εύκολη και πιο φτηνή κυρίως η πρόσβαση με δικονομικές εγγυήσεις επίσης και παρακολούθηση των οικονομικών ε, συναλλαγών και κινήσεων. Ε, επίσης προχωρήσαμε πάρα πολύ στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ε, ευτυχώς το e-justice είναι μια δικτυακή πύλη που θα δει το φως της δημοσιότητας όχι υπό την Ισπανική Προεδρία αρκεί έχει γίνει προεργασία, αλλά ευτυχώς στη Βελγική Προεδρία θα γίνει πραγματικότητα. Ε, τελειώνω, τελειώνω, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να δούμε επίσης τι γίνεται με την εξωτερική δράση κατά το προηγούμενο εξάμεινο ως προς τη δικαιοσύνη. Με τους στρατηγικούς μας εταίρους, τις Ηνωμένες αλλά και με τη Ρωσία. Με τις αντίστοιχες ε, διμερείς συναντήσεις που είχαμε, Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες αυτές και συζητήσαμε ε, θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος τα οποία ανέφερα ήδη και είμαι βέβαιος ότι τα έφερε και ο συνάδελφός μου προηγουμένως Αλφρέντο Ρούμπαλ Κάμπα που είναι αρμόδιος για θέματα εσωτερικών. Hemos, nos hemos dedicado a impulsar... Θέλουμε να προωθήσουμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ελευθεριών και τη συνεργασία σε αστικά και ποινικά θέματα με τη Ρωσία και την Ουκρανία και την Κεντρική Ασία. Άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνω όπως σας είπα και προηγουμένως, αλλά θέλω οπωσδήποτε να αναφερθώ και σε κάτι άλλο κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Και αυτό είναι τα σεμινάρια που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, διοργανώσαμε και έχουν να κάνουν με πάρα πολλά θέματα ε, προτεραιότητας και ουσιαστικά στη φάση της υλοποίησης ε, του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται να σας τα αναφέρω ένα προς ένα γιατί με βέβαιο ότι τα γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Επίσης, γνωρίζετε ότι δουλέψαμε πολύ. Ξέρετε ότι η Ισπανία έχει βαθιά ευρωπαϊκή προσήλωση ριζωμένη στη χώρα και εδώ συνδυάζουμε και τη λογική και το πάθος. Πριν από λίγες μέρες ε, γιορτάσαμε την 25η επέτειο ένταξης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Χάρη στην ευρωπαϊκή μας πορεία έχουμε σταθερότητα και πρόοδο και θα θέλαμε να έχουμε μια ένωση πιο ε, ισχυρή και πιο αλληλέγγυα. Χάρη στις προσπάθειες όλων μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να αισθανόμαστε ε, λογικά ικανοποιημένοι ε, από τον απολογισμό μας. Κάνουμε και σημαντική νομοθεσία και σημαντικό έργο, πάντα εμπνεόμενοι από τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών στην Ευρώπη. Και είμαστε βέβαιοι ότι την ώρα αυτή που έχει έρθει η στιγμή να παραδώσουμε τη σκητάλη στους Βέλγους φίλους μας, μπορούμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον μαζί τους σε αυτό το χώρο, στους νέους τομείς συνεργασίας και συναπόφασης που ορίζει η νέα συνθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Έρχεται τώρα ο γύρος τραπέζης. Σάιμον Μπουσούτη, λέει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσίασή σας και τις εργασίες σας κατά τη διάρκεια του περασμένου εξαμήνου. Έλεγα λοιπόν τώρα που έχετε τη διερμηνία ότι σας ευχαριστώ για όσα κάνατε το τελευταίο εξάμεινο. Θα περιοριστώ σε μία και μόνο παρατηρήση. Η οδηγία για τη μετάφραση και τη διερμηνία και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα αμφισβητήσω το περιεχόμενο των οδηγιών αυτών. Το αντίθετο. Σας συγχαίρω για όσα κάνατε, για να προωθήσετε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες. Τι ήθελα να σας πω, ε, ε κάτι διαδικαστικού χαρακτήρα. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές Ε, στην οδηγία για τη μετάφραση και τη διερμηνία συγκεκριμένα άρχισαν οι εργασίε από την προηγούμενη Προεδρία και συνεχίσατε εσείς, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αρχίσατε εσείς, η Ισπανική Προεδρία, να προωθείτε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας, αλλά υπάρχει κοινή απειλή. Τα κράτη-μέλη ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό φυσικά είναι ένα δικαίωμα των κρατών μελών που αναγνωρίζεται στη συνθήκη. Σε τι έγκυται λοιπόν η δυσκολία. Ο τρόπος χειρισμού των υποθέσεων αυτών. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα πρωτοβουλίες που έχουν για να υποβάλουν νομοθετικές προτάσεις, σε περιπτώσει όμω μόνο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επέμβει. Γιατί τη βασική, το βασικό δικαίωμα, τη βασική πρωτοβουλία ε, ε, για την υποβολή νομοθετικών προτάσεων την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλην όμως και, η και τα κρατημέλη να γνωρίζετε με στη συνθήκη ότι έχουν ένα αντίστοιχο δικαίωμα, αλλά σε περιπτώσει όπου είναι σαφέ ότι δεν θα δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στι δύο αυτέ περιπτώσει ε, ήταν Προφανές ότι ε, θα αναλάμβανε δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε περιέλθει σε αυτήν την αμήχανη κατάσταση όπου ε, το θεσμικό όργανο που λέγεται Κοινοβουλίο έχει πρόταση από το Συμβούλιο και άλλη πρόταση από την Επιτροπή για τα ίδια ζητήματα. για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας εκλιμακώθηκε η ένταση και πραγματικά ε, Ήταν πολύ αμήχανη η κατάσταση και οι εκπρόσωποι της Ισπανικής Προεδρίας μας παρακαλούσαν να υποστηρίξουμε τη δική τους πρόταση, του Συμβουλίου δηλαδή για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την άλλη μας έλεγε αν το κάνετε αυτό θα σας πάμε στο δικαστήριο. Ε, συγγνώμη, αλλά δεν είναι καλές, αυτές, ε, ε, δεν είναι καλές διαθεσμικές σχέσεις αυτές μεγάλο τμήμα της ε, παρουσίασής σας, ε, Υπουργέ, το αφιερώσατε σε αυτές τις ε, διαθεσμικές σχέσεις που αμαυρώθηκαν τρόπον την Πώς βλέπετε αυτό το θέμα Δηλαδή αποκρισταλώνεται αυτό το δικαίωμα των κρατών μελών που να μην αναγνωρίζεται από τη συνθήκη αλλά δεν πρέπει να ασκείται με τρόπο που να δημιουργούνται τέτοιου είδους διαθεσμικές αντιδικίες. Ευχαριστούμε κυρία Ρομέρο Λόπες. Εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρομέρο Λόπες και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω Τον ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό γιατί κατέβαλε μια προσπάθεια ούτως ώστε να μπει ένα λιθαράκι σε αυτό το χώρο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ελευθερίας και δικαιοσύνης διότι αυτά τα βήματα πρώτα τα οποία έχουν σημειωθεί κατά αυτή τη διαδρομή ήταν πάρα πολύ σημαντικά κατά την Προεδρία του. Νομίζω ότι είναι τα θεμέλια για να υπάρξει αυτό ο χώρο. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα αυτά τα θέματα, πολύ δύσκολα τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν αντιμετωπιστεί όπω έπρεπε από αυτό το κοινοβούλιο. Αρχίζει μια καινούργια διαδρομή. Πρόκειται για τη συναπόφαση που δικαιούται να έχει τώρα το κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό σα λέω, πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική διαδρομή, διότι έτσι είναι δυνατόν να έχουμε ε, συνομιλητές για τέτοια θέματα τόσο δύσκολα εγώ θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να διαφωνήσω λίγο με την ερμηνεία του κυρίου Μπουσούτιλ όσον αφορά αυτήν την ε, διαδρομή όσον αφορά την σειρά με την οποία θα παρασχεθεί αυτή η προστασία. Ε, δεν είμαι μόνη συγκέντρια, έχουμε και την κυρία Χιμενστερίλ από την Επιτροπή των Γυναικών και αυτό είναι μια νέα διαδικασία, είναι μια καινοτομία όσον αφορά αυτή την διαδρομή την οποία τώρα κάνουμε. Όσον αφορά τώρα αυτήν την ε, πρωτοβουλία, ξεκινήσαμε όταν στο Κοινοβούλιο ε, ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για τα δικονομικά δικαιώματα όσον αφορά την Επιτροπή μας, η οποία τότε δεν είχε αναλάβει, η Επιτροπή δεν είχε αναλάβει. Είχε αναλάβει μάλλον τα καθηκοντά τη, αλλά δεν λειτουργούσε. Βρισκόμασταν δηλαδή σε κάποια ε, μεταβατική περίοδο μεταξύ της προηγουμένης θητείας και της Επιτροπής που μόλις είχε συγκροτηθεί. Τα δε θα έπρεπε να προσαρμοστούν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και κατά αυτή τη διαδικασία της προσαρμογής στην Λισαβόνα τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να μπορούν να προτείνουν κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά την ποινική συνεργασία. Οπότε, παρά το ότι είναι θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει περισσότερες ε, ε, αρμοδιότητες, είναι απόρρια της συνθήκης της Λισαβόνας το να υπάρχει αρμοδιότητα για τα ποινικά θέματα. Επίσης, όπως γίνεται σε κάποιες ε, χώρες. Ξεκίνησε αυτή όλη η προβληματική για το τι θα γίνει όσον αφορά αυτές τις προτάσεις. Κυρία Ρομέρο, λέει ο Πρόεδρος, συγγνώμη αλλά έχουμε φτάσει στα χρονικά όρια. Ε, μετάφραση, διερμηνία μάλλον. Μας έδωσαν κάποια λεπτά, αλλά απλώς για να μπορέσετε εσείς να ολοκληρώσετε και άλλοι δύο αγορητές και κατόπιν ο Υπουργός να μπορέσει να απαντήσει. Άρα, δεν κυρία Ρομέρο Λόπες, σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να πει η Κομισιόν ότι είναι φύλακα των συνθήκων γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποιες καινούργιες καταστάσεις όπως ας πούμε χθες τα είπαμε με τον κύριο Φαν Ρομπάι όσον αφορά την κοινοτική μέθοδο. Άρα δεν μπορεί να το πει αυτό σου για τις συνθήκες. Γιατί τώρα έχουμε κάποιες καινούργιες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Άρα κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μου είναι η εξή. Όσον αφορά τη Δία. αυτό ε, δεν έχει ρυθμιστεί καθόλου στην Ευρώπη. Τι γίνεται με την οδηγία. Πού θα δοθεί ένας ορισμός αυτού του εγκλήματο. για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πρόοδο. Η Βελική Προεδρία. Η Τρόικα. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι εμεί θα συνεχίσουμε να σα στηρίζουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πορεία. Θα πρέπει η Βελική Προεδρία να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συλλογή δεδομένων ούτως ώστε να δικαιολογηθεί το ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η υπόθεση της προστασίας. Γιατί αυτό είναι το, το μεγάλο πρόβλημα, ότι η Ευρώπη δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι αυτό το έγκλημα που λαμβάνει η χώρα στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια. Κοιτάξτε, δεν φταίει αυτή η τωρινή συζήτηση. Η προηγούμενη κράτησε πάρα πολύ. Επομένως, Ευχαριστούμε την ε, Προεδρία γιατί βοήθησε και στα οικονομικά και σε άλλες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ούτως ώστε να συμμεθούν δήματα Πρόεδρος. Έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε διερμηνή, υπάρχουν χρονικά όρια και μέσα θα δώσουμε σε άλλους δύο το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Χιμένες. Κύριε Μέλλο. ε, σας ευχαριστούμε που για το άρθρο 51 αφορούσε την εισηγήτρια, όχι εισηγήτρια ή ε, στην, σκιώδη εισηγήτρια. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τελικά το θέμα δεν είναι ποιος, ε, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής. Ε, το, το, οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι τα θύματα. Τα θύματα θέλω εγώ να εκπροσωπήσω γιατί όπως ε, προείπαμε τα ε, θύματα πολλές φορές τα ξεχνούμε και εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχω επομένως δουλέψει πάνω σε αυτό, έχω συνομιλήσει με Συμβούλιο, με Επιτροπή, με πολλούς συναδέλφους και τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Ε, είναι αυτό το οποίο θέλω. αυτό με, με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί θέλω να υπάρξει κάποιο είδους φιλόδοξη αντιμετώπιση και θα πρέπει να υπάρχει από όλους αυτή η προστασία. Ε, όχι μόνο τις γυναίκες, όλα τα θύματα. Μιλάτε για κακό μεταχείριση, 95% βέβαια είναι γυναίκες τα θύματα, αλλά θα ήθελα αυτό να σας πω κύριε Υπουργέ, ε, δεν μπορούσα πριν να σας ε, πω, δεν υπήρχε χρόνος, μιλούσατε και για τα θύματα της τρομοκρατίας. Οπότε παρακαλώ και αυτό θα πρέπει να ε, λάβετε υπόψη και θεωρώ ότι έχουμε κάνει λάθη, γι' αυτό βρέθηκαμε σε τόσο δύσκολη θέση. Θα πρέπει επομένω τώρα ε, να γίνει η ρύθμιση σε επίπεδο ποινικού δικαίου. Η ΔΕ Επιτροπή τον Μάρτιο, όπως έχει υποσχεθεί, να κατεβάσει κάποιες προτάσεις που να έχουν σχέση και με το αστικό δίκαιο και να το συνεχίσει και η Βελική Προεδρία. Και εμείς συνεχίζουμε ε, αυτές τις φιλόδοξες προσπαθίες μας. Δεν είναι εύκολο. Η εφαρμογή θα είναι ε, πολύπλοκη και θα υπάρξουν προβλήματα και στο μέλλον όσον αφορά την ε, εφαρμογή αυτή. Να δούμε και εμείς συνενετικά τι θα κάνουμε, πώς θα μπορέσουμε κάτι να κάνουμε για τα θύματα. Νομίζω όμως ότι είναι εφικτό κάτι να κάνουμε. Μην περιστούμε όμως σε ποινικά μέτρα διότι κατά αυτόν τον τρόπο ε, θα υπάρχει πρόβλημα μια που δεν είναι αυτόματη η εφαρμογή των ποινικών μέτρων σε όλες τις χώρες. Δεν θέλω να αφαιρέσω από τους άλλους το, την τιμή της συμμετοχής, αλλά το είπε και ο κ. Μπουσούτιλ και όλοι, ότι θα πρέπει σε αυτή την χρονική στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία, όλα τα θεσμικά όργανα να συνοηθούν για να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι και να βελτιώσουμε την κατάσταση που επικρατεί. Τηλεγραφικός παρακαλώ να είστε, κύριε. Ναι, ναι, πάρα πολύ σύντομα θα είναι. Είπατε ότι τον, ε, από τον Ιανουάριο είπατε ότι θέλετε να είναι πιο φθηνή, πιο γρήγορη η δικαιοσύνη, πιο αποτελεσματική. Ωραία, σύμφωνοι. Τώρα όμως να δούμε τι έγινε όσον αφορά αυτό το κοινοβούλιο. Εγώ είμαι τακτικό μέλος της Νομικής Επιτροπής. Νομίζω ότι έχουμε τώρα ευθύνη με τη συνθήκη της Λισαβόνας ότι θα πρέπει να προχωρήσει τολμηρά το Συμβούλιο και εμείς να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Ο κύριος Υπουργός τώρα έχει το λόγο, θα είμαι σύντομος πρόεδρε. Κύριε Μπουσούτιλ, τι γίνεται με αυτή την διπλή διτή παρουσίαση όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη. Πρέπει να σας πω ότι όλες οι προπαρασκευαστικές πράξεις της Προεδρίας, ακόμα και στην αρχή της Προεδρίας, ε, πρόκειται για αυτές τις πρωτοβουλίες που την κάνουμε με την Επιτροπή Μπαρό που δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα όσον αφορά αυτές τις πρωτοβουλίες. Οπότε τις επεξεργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποτέ δεν είχε πρόβλημα ούτε νομικής βάσης ούτε τίποτα άλλο. Το αντίθετο, το αντίθετο πήγαιναν όλα καλά ε, όσον αφορά τις διαδικασίες ε, δικονομικές εγγυήσεις, ότι δηλαδή η Λισαβόνα δεν ήταν ε, κάτι το οποίο είχε νομιμοποιηθεί εναντί των πολιτών, γιατί θα έπρεπε να αποτελεί κάποια εγγύηση μία και μόνη ερμηνεία σε σχέση με το τι είχε συμφωνηθεί. Και έτσι ε, προχωρούσαμε προς τη λύση αγωνοποίηση, δηλαδή είχαμε αυτήν την, την ε, συναπόφαση με το κοινοβούλιο. Να, τι είπα να πει συναπόφαση. Όχι, δεν είναι πρόκειτο για πρόταση της ε, Κομισιόν που θα οδηγούσε σε εμπλοκή τη διαδικασίας και αποκλεισμό του Κοινοβουλίου. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Αυτά τα είχαμε πει και συμφωνήσει όσον αφορά το να υπάρχει μια τέτοια συνέχεια και να κινηθούμε στη λογική της Λισαβόνας. Να είναι μια ευκαιρία το να εμπλουτίσει τα κείμενα το Κοινοβούλιο. Είτε έχουν ξεκινήσει τα κείμενα από Κομισιόν είτε από το Συμβούλιο. Μια ευκαιρία. Αυτό κάναμε κι εμείς. Όμως με το που άρχισε η καινούργια θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε εξελίξεις μόνο όσον αφορά τα ποινικά θέματα και σας το λέω αυτό γιατί ήταν πολύ στενή η συνεργασία μας. Σε άλλα θέματα πήγαμε πάρα πολύ καλά, όμως μόνο, ε, προχώρησε μόνο η δικαστική ποινική συνεργασία. Γιατί υπήρχε η ποινική συνεργασία. Επομένως, όσο πιο στενή ήταν η ερμηνεία πιο ευρεία συνεργασία. Αυτή ήταν η ουσία της συζήτησης. Το ερώτημα είναι όμως τι κάνουν οι νομικές υπηρεσίες, γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει πρόβλημα στη νομική βάση ή όχι. Και του Συμβουλίου Νομική Υπηρεσία. Εγώ θα πρέπει να κάτσω και να ζυγίσω την αποφασή τους. Αλλά και δική σας η νομική υπηρεσία κανείς δεν είδε κανένα πρόβλημα στην νομική βάση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να δω μία έκθεση ολοκληρωμένη, υπεύθυνη από τη νομική υπηρεσία. Επομένω, δεν μπορώ να συζητήσω τίποτα. Απλώς, απλώς διατύπωσα, αποτύπωσα την πραγματικότητα από τότε που άλλαξε η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρήθηκε ότι είναι λογικό. Αλλαγή του τι θα πει συνεργασία για ποινικά θέματα. Ε, η δε συναπόφαση επέφερε αλλαγές στον τρόπο πολιτική του Κοινοβούλιο και το, και το Συμβούλιο. Γιατί είπαμε ότι καταρχήν η συναπόφαση βελτιώνει τις πρωτοβουλίες. Είτε προέρχονται από την ε, Κομισιόν είτε από το Συμβούλιο. Επομένως δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να μπλοκάρει ε, με νομικά επιχειρήματα κάποιες πρωτοβουλίε του Συμβουλίου. Διότι η δική σας Επιτροπή μπορεί να χτενίζει τα θέματα και να επιλύει τα νομικά θέματα. Α, έτσι ήταν η κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία δεν θα πρέπει να την ε, να, να υπερβάλλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ λογικό να γίνεται αυτό κάθε φορά που έχουμε μια, ένα καινούριο τοπίο θεσμικό, μια καινούργια συνθήκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε θα πρέπει και εγώ, αν επιτρέπετε, να απαντήσω στην κυρία Χιμένες. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ε, ζητήσω συγγνώμη για το λάθος που σας είπα ότι είστε σκιώδης εισηγήτρια. Ναι, ε, δεν πειράζει, ε, γιατί να δούμε ποια είναι η λογική που διέπει αυτή την, αυτόν τον προβληματισμό. Εάν δεν υπήρχαν, ε, αν το έλεγε από την αρχή, δεν πειράζει. Τώρα όμως, ε, ξαφνικά μας λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ε, ας πει, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν το είπε ούτε μια νομική υπηρεσία, ούτε η άλλη. Μα τότε, αν είναι έτσι, τότε τι ωφελεί το να υπάρχει η ερμηνεία υπέρ του θύματος είναι αυτό το οποίο το ξεκινήσαμε στο Συμβούλιο με πρωτοβουλία κάποιων κρατών μελών για να προστατεύσουμε τις Ευρωπαίες. Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγγείλει κάποιες ε, πρωτοβουλίες της, όμως είναι δικαίωμα που κατοικιώνεται από τη συνθήκη. Τα κράτη-μέλη ε, ε, έχουν το δικαίωμα να σταθμίσουν πότε είναι η πιο δόκιμη πρωτοβουλία μπορούν να πάρουν και έχουμε, ε, όχι 18, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης θεώρησαν ότι ε, ήταν το πιο σωστό πολιτικά το να ε, αρχίσει να ισχύει αυτή, αυτό το καθεστώς προστασίας. Θεώρησαν ότι είναι το πιο σωστό να προστατεύσουν τις γυναίκες και ότι ο πλευράς πολιτικής έχει νόημα να υπάρχει το λόγο των γυναικών. Οπότε, ξέρετε, πάνω από 8.000 Ρουμάνες προστατευμένες ε, έχουμε στην, ε, στην Ισπανία. 2.000 ε, Γερμανούς από τις αρχές τις αρμόδιες. Και Βρετανούς πολλούς. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι μόνο ισπανική. Είναι κάτι το οποίο ισχύει σε όλο τον κόσμο. Ε, ανάλογα με το πώς είναι σε κάθε, σε κάθε χώρα. αυτά μπορείτε να κάνετε και να τα ζυγίσετε στην Επιτροπή σας. Να δείτε τι γίνεται όσον αφορά την ελευθερία μετακίνησης με ασφάλεια. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει για τα θύματα, για τους απειλούμενους, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα βίας μεταξύ των δύο φίλων, είναι γενικότερο θέμα του ευρωπαϊκού χώρου. Αυτή είναι η γραμμή πλεύσης και το πνεύμα που ακολουθήσαμε. Τέλος, για την κυρία Ρομέρο θα πρέπει να πω ότι η Βελγική Προεδρία από την πρώτη μέρα δεσμεύτηκε να ακολουθήσει την ίδια γραμμή πλεύσης Γι' αυτό και εμείς είμαι θα ότι πρόκειται να συνεχίσει αυτό το έργο και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η δική σας δουλειά εδώ πρόκειται να είναι κάτι το αξιόλογο, να υπάρξουν δικονομικές εγγυήσεις για να δούμε τι θα γίνει, πώς θα δουλέψουμε τώρα με την ε, συνήθεια αγώνας και ε, να υπάρξει ένα απτό αποτέλεσμα το οποίο και να το εκτιμήσουν οι Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την προσπάθεια που κάνετε να είστε σύντομος. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες ε, τόσο πυκνό και φορτωμένο πρωινό σήμερα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους διερμηνείς που έκαναν υπέρβαση ε, ωραρίου τους κατά ένα τέταρτο της ώρας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.